Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι ορισμένοι πρέπει να πάτε και σε άλλες επιτροπές και σε άλλες εκδηλώσεις. Μου ζητήθηκε λοιπόν να ξεκινήσουμε γρήγορα. Αφήστε, παρακαλώ πολύ, δεν είμαστε και τόσοι πολλοί, επομένω φαντάζομαι ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και για όλα τα ζητήματα. Η Αντιπρόεδρε είναι εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με το σημείο 14 τη ημερησία διάταξη. Συμφωνία συνεργασία για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Ο Φρανκ Αγγέλ είναι ο εισηγητή μα. Δυστυχώ όμω δεν μπορεί να είναι παρόν. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 2. Ας περιμένουμε λιγάκι. Αλλά όχι πάρα πολύ. Αν εσύ μπορείς να καθίσεις γρήγορα, βγάλε και την κάρτα σου. Okay. And then I'm going... You ready? Uh, the, vote, the vote is closed. Απορρίπτεται. Λίγοι είναι οι συνάδελφοι πάντως. Ε, δεν είναι και τόσο νωρί. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία 4. Υπέρ. 8. Διορθώνει η Πρόεδρος. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, λέει η Πρόεδρος, αλλά θα ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Και όντως απορρίπτεται. Περνάμε συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται 14 υπέρ, ουδής κατά και τρεις αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Απόντα Φρανκ Έγγελ. Περνάμε τώρα στην διαδικασία σύμφωνη γνώμης, συγκατάθεσης, ε, ναι ή όχι ουσιαστικά λέμε εδώ πέρα, με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε, δεν υπάρχουν τροπολογίε. Ονομαστική κλίση ηλεκτρονικά όσον αφορά τη συμφωνία με το Αφγανιστάν, να ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Και δίδεται η συγκατάθεση 15 υπέρ, ουδής κατά και δύο αποχές. Πολύ ωραία. Περνάμε έτσι στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Ειδικέ διατάξεις που διέπουν το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα Interreg, το οποίο θα ψηφίσουμε. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η συντάκτρια γνωμοδότηση είναι η Ελένη Θεοχάρου. Ελένη, θέλει να πάρει το λόγο να πει κάτι το ψηφίσουμε, όχι. Άρα μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσω. 13. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 73. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόκειται νομοθετική πρόθεση. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν όλες ξεχωριστά. 17 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 76. Άρχεται η ψηφοφορία. δεν έχετε την κάρτα σας, μπορεί να σας τη φέρει κάποιος, μπορείτε να στείλετε κάποιον να σας τη φέρει, ενδεχομένως κάποιος από το προσωπικό. Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Προσθέτουμε και τη δική σας την ψήφα, αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ψηφίζετε υπέρ ή κατά, Πρόεδρος. Πολύ ωραία, πέρας. Γκρίνεται, 9 υπέρ, 8 κατά. Μπορείτε να φέρετε την κάρτα σας ή κάποιος να σας τη φέρει τουλάχιστον. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν κάποιο δεν μπορούσε να ψάξει που βρίσκεται η κάρτα σα και να σα τη φέρει, θα βοηθούσε. Okay. Μάλιστα, εντάξει.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 Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά αποχές. Καταπίπτει 29, σας ζητώ συγγνώμη λέει Πρόεδρος, γιατί εγκρίθηκε 85. Περνάμε έτσι στην 86 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 86, άρχεται η ψηφοφορία. Ήταν σαφές, πέρας, ήταν σαφές, σας ζητώ συγγνώμη λέει Πρόεδρος. 4 υπέρ 15 κατά καμία αποχή.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 Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 39 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρασε. 12 υπέρ και 8 κατά. Άρα εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση μάλλον για την τροπολογία 89, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται 11 υπέρ και 9 κατά. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 90 ψηφίζουμε παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 10 υπέρ και 9 κατά 48 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία, αλλά σας ελέγξουμε ηλεκτρονικά και την 48 άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πολύ ωραία, πέρας. Και όντως εγκρίνεται 11 υπέρ, 9 κατά. 49 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αρκετέ σελίδε ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι. 51 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 91, άρχιτη ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρα. 10 υπέρ και 10 κατά. Απορρίπτεται λοιπόν. 92 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά 93 από την αρχή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 96. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 10 υπέρ, 9 κατά και εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Όχι, όχι, είχαμε έναν που ψήφισε υπέρ χωρίς να έχει κάρτα και προσθέσαμε την ψήφο του. Το είχαμε πει αυτό από την αρχή. Έχει συμβεί και το αντίστροφο. Εντάξει. Σε ορισμένες ψηφοφορίες είχε συμβεί αυτό και από την πλευρά του ΕΛΚ. Εντάξει. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις τολικές σκέψεις. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 56. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρας. 13 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. 57 υπέρ. Κατά. αποχε απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν για τροπολογία 58. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 13 υπέρ και 7 κατά. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 59 καταπίπτει, η 5 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελευταία σελίδα. 67 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 67 άρχιτη ψηφοφορία. Όχι είναι σαφές τώρα λέει η πρόεδρος. Σε το συγγνώμη. πέρασε σε κάθε περίπτωση. Σαφώς απορρίπτεται. 4 υπέρ 15 κατά. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Η 12 καταπίπτει μάλλον. 69 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 69. Άρτη ψηφοφορία. 7 υπέρ, 11 κατά και απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ετολικές αναφορές 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική τώρα ψηφοφορία, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ, ουδής κατά και καμία αποχή εγκρίνεται. Ελένη, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την καταπληκτική εργασία που κάνατε. Ψηφίσουμε τώρα την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Είναι μια γνωμοδότηση που θα πάει στην Υποπιτροπή ΣΕΝΤΕ δεν γνωμοδοτούμε επίσημα για το ζήτημα αυτό, αλλά με τους συντονιστές αποφασίσαμε ότι θα καταθέσουμε τροπολογίες όπου υπάρχει ευρεία συνένεση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. G. Υπέρ. 3. Μάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται με 16 ψήφους υπέρ, ουδής κατά και δύο αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ. That concludes votes, colleagues. So thank you very much. Πληρώθηκαν ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. κύριος Ρούμπικ, ε, Πάουλ, έχεις το λόγο. Ήθελα να πω ότι η ψηφοφορία σχετικά με το Αφγανιστάν, εγώ δεν ψήφισα γιατί είχα προβλήματα με την έκθεση. Αυτή ήμουν παρόν, αλλά δεν συμφωνούσα με κάποιε από τι διατάξει του πρωτοκόλλου αυτού. Πολύ ωραία θα περάσει αυτό στα πρακτικά, λέει η Πρόεδρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και είστε εδώ, Χθε είχαμε ελάχιστου συναδέλφου στην Επιτροπή μα. Θα ήθελα απλώ να σα πω ότι χθε συζητήσαμε το πρωτόκολλο αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Bogdan Βέντεμ. Το ΕΛΚ μπορεί να με ακούσει, παρακαλώ πολύ. Κρίστιαν, έλεγα ότι χθε ήταν ελάχιστοι συνάδελφοι εδώ. Αλλά στείλαμε τι ευχαριστίε μα στον Bogdan Βένταμ για το πρωτόκολλο τη Επιτροπή αυτή. Για όλη την εργασία που έχει κάνει με του υπόλοιπου συντονιστέ. Ήθελα αυτό να το πω παρουσία των υπολείπων συναδέλφων σήμερα και ευχαριστήσαμε επίσης και τη Βαλερή η οποία φεύγει. Ολοκληρώθηκαν ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ. Okay, colleagues, we're moving now to item 18. Προχωράμε στο άρθρο 18, στο σημείο 18 μάλλον. Που είναι τα αποτελέσματα την ειδική ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης στην Βολιβία, 18 με 20 Σεπτεμβρίου. Η Ελένη Θοχάρους, ο Άγουστιν Διεντεμέρα ήταν μαζί είναι παρόντες δύο από αυτούς που επισκέφτηκαν ε, τη Βολιβία. Πώς έμαθα από το προσωπικό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αποστολή. Είχατε συναντήσεις με υψηλά ειστάμενους μισή μέρα με τον πρόεδρο Εύω Μοράλες σε ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα όπου ε, επισκεφτήκατε ε, χωράφια καλλιέργειας κόκας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Βολιβιανή κυβέρνηση. Καθώς λοιπόν αναφερόμαστε στην ε, αποστολή, να πούμε ότι έλαβε χώρα στη Λαπάς. Θα δώσω το λόγο στην Ελένη Θεοχάρους επικεφαλής της αποστολής για να μας πει περισσότερα για την αποστολή και να μας ενημερώσει αν πρέπει να υπάρξει κάποιο φόλο από την πλευρά της Επιτροπής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη που συμμετείχαν στην αποστολή αυτή, τον Ογκαστίν Τεμέρα και τον κύριο Φουτζουλίτσα και επίσης όποιους είχαν την πρόθεση να έρθουν αλλά δεν μπόρεσαν ε, λόγω κάποιου απρόβλεπτου προβλήματος. Να ευχαριστώ την Ιωάννα, την το Χάρη, όλο το προσωπικό που προετοίμασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστόλη μας. Επίσης, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Λαπάθ, τον Λεών δεν μπορώ να θυμηθώ το επεισόδιο αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει όμως τον γνωρίζετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σκοπός της αποστολής μας ήταν να παρακολουθήσουμε την ε, εξέλιξη της συνεργασίας στις τρεις, ε, τομεί τρεις τομείς προτεραιότητας, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνη και καταπολέμηση της διαφθοράς, την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών και και την ε, χρηστή διαχείριση των υδάτων. Όσον αφορά αυτές τις τρεις ε, τους τομείς ε, εστίασης, επιλέχθηκαν και είναι πλήρως αυθυγραμμισμένοι με τις προτεραιότητες που έχει η Βολιβία, όπως είναι η ατζέντα πατριώτικα του 2020-2025 και σύμφωνα με το ε, πλανο ε, κοινωνικο ε, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 2016 με 2020. Υπάρχει ένας μηχανισμός συνεργασίας που παρέχει 281 εκατομμύρια ευρώ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Επίσης, επαφελούνται και από άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τη διάρκεια της επίσκεψής μας συναντηθήκαμε με τέσσερις ε, υπουργού, έναν υφυπουργό, ε, αρχηγού επικεφαλή αποστολών, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με το Εθνικό ε, Συμβούλιο για την Καταπολέμηση των Παράνομων Ναρκωτικών και την Ειδική Δύναμη για την καταπολέμηση ε, των Ναρκωτικών και την Ειδική Επιτροπή για την ε, Παιδική Εργασία. Επίσης, συναντήκαμε με τον πρόεδρο Ιβο Μοράλες. Πετάξαμε με ελικόπτερο πάνω από χωράφια τα οποία, ε, στα οποία η καλλιέργεια είχε μετατραπεί από καλλιέργεια κόκα σε παραγωγή φρούτων. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σας ευχαριστήσω όλους που συνεργαστήκατε για την προετοιμασία της αποστολής και συγκεκριμένα την Ιωάννα. Θα προσπαθήσω να προσπεράσω τις ε, λεπτομέρειες και να σας δώσω κάποια βασικά σημεία της αποστολής μας. Ο Υπουργός ε, Ψηδιασμού και ο Υπουργός Εξωτερικών ε, σημείωσαν ότι συμπίπτουν οι προτεραιότητές μας. Ο κύριος Πάρη, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών, είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, ο οποίος σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό θεωρώ ότι θα είναι καλός πρόεδρος στο μέλλον για αυτή τη χώρα. Ο κύριος Μπράντον Νόγια αξιολόγησε την ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εξαιρετική στο, στη διαχείριση του νερού, καλή στον τομέα της διακίνησης των νοικοτικών και ότι ε, επιδέχεται βελτίωση στον τομέα της ε, δικαιοσύνης. Η φτώχεια στην ε, Βολιβία έχει αλλάξει, έχει μετωπιστεί τα τελευταία χρόνια εξαιτία τη αστικοποίηση και υπάρχουν θέματα στον τομέα τη υγεία και στι εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια. Όσον αφορά ε, τις εξωτερικές υποθέσεις, ο κύριος Πάρης σημείωσε πολλούς τομείς σύγκλησης μεταξύ Βολιβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πώς μπορεί να βελτιωθεί ο διάλογος μεταξύ μας και να λαμβάνει χώρα σε ε, ίση βάση. Επίσης να υπάρχει αμοιβαιότητα και η ενδεχόμενη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου ε, είναι θέματα για τα οποία θα θέλουμε να συζητήσουμε και πιο εντατικά. Ο Άρκη Ζακονέτα. Σχεδόν όλοι οι υπουργοί έχουν ελληνικά ονόματα. Αναγνώρισε ότι το σύστημα δικαιοσύνης χρειάζεται βελτίωση. Μια από τις βασικές προκλήσεις είναι η ενίσχυση της ε, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης γιατί δεν υπάρχει επαρκής προϋπολογισμός που προ... και αυτό προκαλεί και καθυστερήσει στο σύστημα της δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Υπεύθυνος για το Νερό, κύριος Ορτούνιο, συμπεριέλαβε στο διάλογο πολλά θέματα όπως ε, η ενεργειακή επάρκεια, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και επίσης αναφέρθηκε σε εσωτερικούς εκτοπισμούς πληθυσμών εξαιτία της κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει η Βολιβία να διαφοροποιήσει τις ε, πηγές ενέργειας και ε, να μελετήσει και ενδεχόμενες εξαγωγές στην περιοχή. Επίσης αναφερθήκαμε σε, στα σχετικά θέματα της πρόσβασης στο νερό και στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Όσον αφορά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Εύω Μοράλες, είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την περιοχή Τσαπάρε, στην περιοχή της Κοτσαμπάμπα. Η άλλη βασική περιοχή παραγωγής κόκα της Βολιβίας. Η άλλη περιοχή είναι τη Γιούγκα. Ο κύριος Μοράλ, τόνισε ότι η Βολιβία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο με το πακέτο συμφωνία με, την, ε, με τις ΗΠΑ. Θεωρεί ότι είναι επιτυχημένη η προσπάθειά τους να μειώσουν την καλλιέργεια της Κόκα, ε, την οποία κατάφεραν να μειώσουν από 30.000 σε 20.000 εκτάρια. Η καλλιέργεια της Κόκα είναι μια παραδοσιακή δραστηριότητα ήταν περιορισμένη για να υπάρχει επάρκεια στον παραδοσιακό τοπικό τομέα. Πριν από 20 χρόνια, στην περιοχή που επισκεφτήκαμε υπήρχε μόνο παραγωγή κόκα, τώρα υπάρχουν ε, μπανάνες, ε, μάγκο και άλλα φρούτα. Η συνεργασία με τις ε, ενώσεις εργαζομένων κατάφερε να μειώσει την ποσότητα αυτή και να δημιουργήσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης. Επίσης τα ποσοστά φτώχειας έχουν πέσει και η ακραία η φτώχεια έχει πέσει από 37% στο 17% με περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους να φτάνουν ένα ε, μέσο επίπεδο εισοδήματος. Όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, παράνομης κυκλοφορίας ναρκωτικών, κατάφεραν τα τελευταία 20 χρόνια με διάφορα προγράμματα να έχουν κάποια επιτυχία. Η καλλιέργεια γινόταν για εσωτερική παραγωγή σε 22.000 εκτάρια και γι' αυτό ο ΠΟΕ προσπάθησε να νομιμοποιήσει ε, την χρήση για παραδοσικούς σκοπούς αν αυτό το σχέδιο του ΠΟΕ δεν πετύχει, τότε θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η καλλιέργεια. Επίσης υπάρχουν προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και από άλλους δωρητές. Ο επιτυχής κοινό προγραμματισμός ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα γιατί ε, βοήθησε στην καλύτερη χρήση του προπολογισμού. Ωστόσο το νερό ε, υγιεινή είναι βασικά θέματα. Θέματα για τη Βολιβία. Επίση, θέματα τα οποία πρέπει να μελετηθούν είναι οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, τα οποία θα πρέπει να υπάρξει και ισχυρότερη διεθνή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεισφορά τη κρίθηκε είναι πολύ σημαντική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την γενικότερη υποστήριξη στους φορείς της ε, κοινωνίας των πολιτών και για την οικοδόμηση ικανοτήτων στις ε, τοπικές αρχές. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει για το πολιτικό τοπίο και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία ε, κατά τη διάρκεια διαφόρων συναντήσεων που είχαμε με επικεφαλής αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και μέλη και βουλευτές, τον Κονζάλο Μπαριάντος και τον Ντουίν Ροντρίγκερς, Επίσης είχαμε ανταλλαγή ε, απόψεων με μη κυβερνητικέ οργανώσεις που απασχολούνται με των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε η μερική εφαρμογή νέας νομοθεσίας. Η έλλειψη ε, ανεξαρτησίας του τομέα της δικαιοσύνης ε, δημιουργεί συνθήκες για ατιμορρησία. Τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών, καθώς και η βία ενάντια στα παιδιά και η παιδική εργασία είναι τομείς στους οποίους θα πρέπει να ε, επεκταθούν και να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Συνειδηθήκαμε επίσης ε, με την ε, Ένωση για τα παιδιά και νέους εργαζομένους. Υπάρχει σχετική νομοθεσία του 2014 για την παιδική εργασία που τους δίνει τη δυνατότητα να δουλεύουν, να εργάζονται σε ένα προστατευμένο πλαίσιο ώστε να υποστηρίζουν τις οικογένειες τους, κάτι που συμβαίνει από μικρή ηλικία. Αυτό φυσικά είναι ενάντια στα βασικά δικαιώματα των παιδιών, αλλά όπως και να έχει, αυτό που ζήτησαν από εμάς όσον αφορά τη βία εναντία στις γυναίκες, ε, οι γυναίκες έχουν μικρή συμμετοχή στην πολιτική, ε, είναι θύματα διάκρισης και το μήνυμα ήταν σαφές. Η Βολιβία βασίζεται για την ανάπτυξή της σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν ε, με τις ε, πολιτισμικές αλλαγές, την, ε, το σεβασμό στο φίλο και τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό το θέμα αναφέρθηκε και στο πλαίσιο του κέντρου για την πρόθεση της γυναίκας, αλλά Αγκοστίν ασχοληθεί πιο πολύ με αυτόν, οπότε θα δώσω το λόγο αργότερα. Ε, επίσης επισκεφτήκαμε ε, την κοινότητα της Φουαρίνα για την βελτίωση της, ε, των υδάτων στην Λίμνη Τιτικάκα και την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ήταν δύσκολο να αναπνεύσουμε και να κινηθούμε. μας εντυπωσίασαν οι μέθοδοι καθαρισμού του νερού βλέπουμε ότι υπήρξε, υπήρξαν θέματα διαχείρισης ε, στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για να ολοκληρώσουμε, κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής είδαμε ότι υπάρχει ευθυγράμμιση με τις εθνικές προ, ε, προτεραιότητες και όσον αφορά το follow-up Τρει από τους βασικού τομεί συνεργασία, η καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών και η διαχείριση των υδάτων είναι πολύ πιο ε, υψηλά στο θέμα της ε, αντιμετώπισης και εφαρμογή. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά όμω για, την, ε, για τον τομέα των υδάτων καθώς ο υψηλός ρυθμός της αστικοποίησης δυσχεραίνει την κατάσταση. Όσον αφορά το τρίτο τομέα εστίαση, στην καταπολέμηση τη φθορά, η συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να, ε, να ψηθούν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για να προωθηθούν τα προγράμματα μεταρρύθμισης τη δικαιοσύνης. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους μου να πάρουν το λόγο για επιπρόσθετα σχόλια και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, μας έδωσαν την ευκαιρία να υλοποιήσουμε αυτή την εξαιρετική αποστολή. Μία μικρή σημείωση που αφορά και ε, τον καθαρισμό του ύδατος στην λίμνη Τιτικάκα θα μπορούσα να πω ότι με πολύ λίγους πόρους μπορούν να ε, καθαρίζουν τον νερό χρησιμοποιώντα φυσικά φαινόμενα όπω είναι η όσμωση ή η βαρύτητα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώ να το κάνουν αυτό. Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Κάτω από 35.000 ευρώ. Και με αυτά είχαν δυνατότητα ετησίω να παρέχουν στην πόλη καθαρό νερό. Επίση εντυπωσιακό είναι ότι, ότι στο υψόμετρο των 4.000 μέτρων το νερό ήταν πολύ βρώμικο. Και το νερό της λίμνης και από τα πηγάδια εξαιτίας της έλλειψης ε, κατάλληλων συστημάτων. Ε, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Κυρία Πρόεδρε, μπορείτε να δώσετε το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστούμε, Ελένη, για αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες οι άλλοι δύο συνάδελφοι που... Ο κύριος θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δύσκολο είναι να προσθέσω κάτι γιατί ήταν πολύ αναλυτική η παρουσίαση της Ελένης. Ήθελε και εγώ να τονίσω ότι επέδειξε σημαντικό επαγγελματισμό η επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας, η κυρία Θεοχάρους. θα έλεγα ότι αυτή η επίσκεψη μας έδειξε ποιος, ποια είναι η παγκόσμια επιρροή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί τη Βολιβία, μια χώρα τόσο, που βρίσκεται τόσο μακριά, που έχει σήμερα πια ένα διαφορετικό πολιτικό σύστημα με πολλές δυσκολίες, ε, τα γνωρίζετε, με καταγγελίες για τις εκλογές κτλ. λοιπά. Εν τέλει όμως βλέπουμε ότι έτσι ασκεί την επιρροή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι υποστηρίζει τους λαούς που προσπαθούν να κατακτήσουν πραγματική δημοκρατία. Εάν δεν ε, συμμετείχαμε, δεν ε, εμπλεκόμασταν στην υποστήριξη μια χώρα όπως η Βολιβία θα ήταν δύσκολο να την επηρεάζουμε. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχίσουμε για να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν στο τέλος τη δρόμο της δημοκρατίας, να βελτιώσουν την κατάσταση με τα δικαιώματα των πολιτών, την ελευθερία του τύπου, που δεν είναι και η καλύτερη ε, κατάσταση στη χώρα αυτή. Όλα αυτά έχουν σχέση με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, την αιρεσιμότητα που θέτουμε. Γνωρίζετε ότι είναι πολύ επιφυλακτική, προσεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά. Ίσως θα έπρεπε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, στην προσπάθειά μας να επηρεάσουμε χώρες όπως τη Βολιβία προς την κατεύθυνση της δημοκρατίας. Γιατί στις χώρες αυτές βλέπουμε να υπάρχουν νέοι που να του απασχολούν τα θέματα αυτά. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ισότητα των δύο φύλων, πολύ σημαντικό για τη βιολεβία, που έχει παραδόσεις που ίσως να πρέπει να αλλάξουν, παραδόσεις επίσης των αυτοχθόνων πληθυσμών που ζουν εκεί, Είναι επίσης σημαντικό ότι είχαμε συναντήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία αποδίδει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την αποστολή του. Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελε κάποιος άλλος συνάδελφος να ρωτήσει. εκεί. Ευχαριστώ για την ε, έκθεση αυτή, Ελένη. Τον προηγούμενο χρόνο με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Κυμάτων βρεθήκαμε στη Βολιβία και πρέπει να πω ότι η εικόνα που μας παρουσιάσαν δεν ήταν και τόσο θετική. Όσον αφορά τον πρόεδρο Μοράλες, φαίνεται ότι παίρνει δικτατορικές διαστάσεις Όταν ήμασταν εκεί υπήρχαν, υπήρξαν δύο μεγάλες διαδηλώσεις στην ε, κοινότητα των Ιθαγενών. Έτσι δεν μπορούσαμε να ε, συναντηθούμε με τους αρμόδιους υπουργούς του Υπουργείου Συντερικών συγκεκριμένα γιατί είχαν μπλοκάρει την είσοδο στα Υπουργεία οι διαδηλωτές Επίση, αυτό που κάνουμε τη Βολιβία είναι να δίνουμε χρηματική υποστήριξη για τη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων για την βελτίωση της ε, παροχής νερού ε, στις αγροτικές περιοχές. Όμως πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα project γίνονται στις περιοχές στις από τις οποίες κατάγεται ο πρόεδρος Μοράλες η τρίτη μεγαλύτερη φυλή συγκεκριμένα από τους αδεγενείς της Βολιβίας. Είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και μια φυλακή. που θα έπρεπε να έχει χωρητικότητα 800 άτομα. Σε ένα παλιό μοναστήρι υπήρξε αυτοδίκηση. Ε, των ε, κρατουμένων οι οποίοι ουσιαστικά φροντίζονται από συγγενείς. Ήταν απερίγραπτες στις συνθήκες μέσα εκεί. Επίσης και στο θέμα της εργασίας των παιδιών συναντηθήκαμε με την ε, Ένωση, τη σχετική οι οποίοι μας παρουσίασαν ότι η νέα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα εργασία στα παιδιά και είναι ουσιαστικά ε, θετική, γιατί θέτει κάποια θεμέλια. Η προσέγγιση του Μοράλη στη Βενεζουέλα, την Κούβα και την Βόρεια Κορέα φάνηκε όταν είχε προσωρινή ε, έδρα στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Βολιβία. Εξελέγει ως πρώτος πρόεδρος από... με καταγωγή από ηθαγενή φιλή. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια μονοπλευρή ε, προσέγγιση στο βορρά. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ε, μιας περιοχής ε, τροπικού δάσους όπου θέλουν να φτιάξουν δρόμους ενάντια στη βούληση των Ιθαγενών, των ντόπιων για να υπάρξει σύνδεση με την Βραζιλία. Επίσης παράλληλα Ε, που έχει να κάνει με τον χαμένο πόλεμο του 19ου αιώνα που κατέστησε αδύνατη την πρόσβαση της Βολιβίας στον Ειρηνικό ωκεανό, μια περιοχή που προηγουμένως ανήκει στη Βολιβία. Επίσης, και γι' αυτό σε εκείνες τις περιοχές ε, λαμβάνει χώρα προπαγάνδα για να υπάρξει μια αναθεώρηση ώστε να επιτραπεί αυτή η δίωδος ε, στον Ειρηνικό ωκεανό για τη Βολιβία. Μία από τις διαδηλώσει που μπλόκαρε το Υπουργείο Οικονομικών ρώτησα τους διαδηλωτές γιατί διαδηλώνουν και ήταν κυρίως θαγενείς γυναίκες που κερδίζουν το, τα προστοζήν μέσω α, ρουχισμού που έρχεται δωρεάν από την Αμερική πουλάνε ουσιαστικά μεταχειρισμένα ρούχα στην αγορά. Όμως επειδή θέλει να κόψει την πρόσβαση στην Αμερική, ο Μοράλες ε, παρεμπόδισε ουσιαστικά την πρόσβαση των γυναικών αυτό στα ίδια αυτά, στα μεταχειρισμένα ρούχα, κάτι που για αυτές ε, αποτελεί καταστροφή της ε, εργασίας τους. Όσον αυτά που είπε ο συνάδελφος, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στην περιοχή, θα πρέπει όμως παράλληλα να σιγουρευτούμε ότι τα οικονομική ενίσχυση ε, που παρέχουμε δεν χρησιμοποιείται πολιτικά μονόπλευρα από τον ε, Πρόεδρο. Αλλά θα πρέπει να επωφελούνται όλοι ένα από τα βασικά φαγητά είναι η κοινόα, η οποία καλλιεργείται εντατικά. Είναι ένα φαγητό το οποίο είναι πολύ ε, δημοφιλές στους ε, vegan και γι' αυτό έχει ανέβει πάρα πολύ η τιμή του και προορίζεται κυρίως για εξαγωγές και έχει καταστεί πάρα πολύ ακριβό για τους ε, ντόπιους πληθυσμούς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο που είπατε. Αν σκεφτεί κανείς πόσες εκστρατείε γίνονται εδώ για το πόσο για τα ωφέλη για την υγεία του που υποτίθεται πως έχει Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις στην αγορά. Ελένη, φαντάζομαι θα θέλατε να λάβετε το λόγο. Υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Υπάρχει επίσης και εκπρόσωπος της ε, Πρεσβείας της Βολιβίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελένη, θέλατε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ με τις ε, απόψεις του συναδέλφου Τζέλερ ε, έχει δίκαιο να αγωνιά όπως αγωνιούμε και εμείς για τον τρόπο διάθεσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, στην Βολιβία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε πάει. Ε, ωστόσο θα έλεγα ότι έχει παρατηρηθεί μια σημαντική πρόοδος έστω και αν αυτή βγαίνει μέσα από τις παραδοξότητες αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου του Ιβο Μοράλες ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής και αυτό είναι το ε, το εκπληκτικό σε αυτή τη χώρα ε, και γιατί προέρχεται από μια από τις ε, φυλές της indigenous της, της Βολιβίας αλλά και γιατί έχει μια απλότητα με την οποία προσεγγίζει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Για παράδειγμα είναι ποδοσφαιριστής μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρικής ομάδας και παίζει τακτικά παρά τα 59 του τόσα χρόνια πόσο μας είπε. Ε, Βεβαίω υπάρχουν πολλά προβλήματα. Η αγωνία μα για την κόκα είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί οι ειδικοί εκεί πέρα τόσο από μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από μέρου ε, τη αντιπολίτευση και των experts μα είπαν ότι η κόκα που καταναλώνουν οι ηθαγενεί για καθημερινή χρήση, τα φύλλα είναι πολύ πιο καλά από αυτά που έρχονται από το Περού και συνεπώ Αυτά που παράγονται τοπικά ως επιτοπλίστων μετατρέπονται σε κάτι άλλο που δεν μας είναι και πολύ ε, ευχάριστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο ρόλος της αποστολής μας δεν ήταν να γίνουμε detectives και αστυνομικοί. Απλώς επισημαίνουμε και σε κάποιο σημείο της ε, παρουσίασης μου το είπα. Όπως είπα και αρκετά συγκεκαλυμμένα κατά κάποιον τρόπο ή αν θέλετε αποστρογγυλωμένα από αυτά που είπε και ο κύριος ε, Τζέλερ. Τώρα, όσον αφορά τις φυλακές, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καταγγελίες ότι υπάρχουν φυλακές ακόμα και στην δική μου την χώρα στην Κύπρο που είναι ε, υπερπλήρης και ε, δεν θα περίμενε κανείς κάτι καλύτερο σε μια υποανάπτυχτη χώρα της Λατινικής Αμερικής όπως ε, και σε άλλες ε, ανάλογες περιοχές. Σήμερα γίνεται στην Λαπάς το συνέδριο, το High Level Symposium για την Ειρήνη και καλό θα ήταν και φαντάζομαι ότι και εκείνοι θα επιχειρήσουν να κάνουν το ίδιο να μην διαφυλάξουμε αυτή, να αυτή την προσπάθεια για να υπάρξει ένας συντονισμός και μια συνεργασία των χωρών της Λατινικής Αμερικής προς την κατεύθυνση της ε, ειρηνικής συνύπαρξης, της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και κυρίως της, ε, της φτώχειας. Ε, το πρόβλημα της έλλειψης συστημάτων αποχέτευσης είναι ε, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και το οποίο ταλανίζει όχι μόνο την ε, δυνατότητα να έχουν καθαρό νερό αλλά και τα νοσοκομεία τους με καθημερινές λοιμώξεις και παθήσεις που δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν. Τώρα, όσον αφορά το conflict για το access στον ειρηνικό Όντως το 2004 το 1904 η Βολιβία έχασε τον πόλεμο από την Αργεντινή και δυστυχώς για την ίδια υπέγραψε τη συμφωνία με την οποία παραχωρούσε την, τα εδάφη με τα οποία επικοινωνούσε η Βολιβία με τον Ειρηνικό. Η Χιλή έχασε και την δίκη στο δικαστήριο των, το Διεθνές Δικαστήριο πριν από ένα μήνα βγήκε η απόφαση και μας κοινοποιήθηκε. Ε, και συνεπώς δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να απαιτεί πρόσβαση στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο η Χιλή έχει προσφερθεί να δώσει ζώνη ελευθέρου εμπορίου σε λιμάνι στις βόρειες ακτές της και τη δυνατότητα ε, σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης με την Βολιβία που είναι μικρή ούτω ώστε στο τέλος να υπάρχει μια συνεργασία καλής γειτονίας όπως γίνεται σε πολλά άλλα μέρη της Ευρώπης όπως γίνεται στο Καλίνιγκρατ, όπως γίνεται στην Κροατία με την ε, Σλοβενία και ε, σε, πολλά, σε πολλές άλλες ε, περιοχές. Νομίζω ότι αν η Βολιβία δείξει καλή συμπεριφορά σε αυτό το θέμα δεν θα της αποστερηθεί η πρόσβαση στον Ειρηνικό ωκεανό. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, και εμείς ευχαριστούμε. Έχω τον κύριο Αλφόνσο Χουίτ από την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακή Συνεργασία τη Επιτροπή και εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Θέλετε να προσθέσετε κάτι ιδιαίτερα για τον πολιτικό διάλογο στη Λαπά που ξεκινά σήμερα. Από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ την αντιπροσωπεία σας που επισκέφθηκε την Βολιβία Νομίζω συμμεριζόμαστε τις παρατηρήσεις που και τα συμπεράσματα. Πράγματι είναι ακόμα αναπτυσσόμενη χώρα η Βολιβία. Ε, είναι ε, μια χώρα τυπική της ε, Νότιας Αμερικής θα έλεγα. Και αυτό που κάνουμε είναι να προωθήσουμε την καταπολέμηση της φτώχειας και την πρόοδο σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Έχουμε το 2014 επιλέξει κάποιους τομείς, ανάμεσα σε αυτούς είναι και η διαχείριση των υδάτων, που θεωρούμε σημαντικούς και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ε, αποτελεσματική σε αυτούς τους τομείς η συνεργασία. Σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η συνεργασία δεν ήταν αποτελεσματική, δεν έχουμε επιτύχει αυτό που θα θέλαμε. Γι' αυτό αυτό το, αυτή η έκκληση για περισσότερη χρηματοδότηση στα συμπεράσματα θα έλεγα ότι δεν είναι σωστή, γιατί τα 50 εκατομμύρια που είχαμε τα πρώτα 5 χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, συνεχίζουν δηλαδή να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα στη συνεργασία με αυτή την χώρα. Και όπως είπε και ο κύριος Τσέλα, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της ανάπτυξης που μας απασχολούν, υπάρχουν και τα ζητήματα των πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε την τέταρτη πια θητεία του κυρίου Μοράλες, ε, παρά το γεγονό ότι σε διποψήφισμα ο λαό τη Βολιβίας είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να επανεκλεγεί, βρήκε ένα τρόπο μέσω του συνταγματικού δικαστηρίου να ξανά υποψηφιότητα. Επομένω, ο διάλογο μα δεν εστιάζεται μόνο στην κοινωνικο-οικονομική πρόοδο, όπου είχαμε πρόοδο. Προσπαθούμε ταυτόχρονα να εξετάσουμε και τι πολιτικέ εξελίξει συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων ορισμένων ε, μειονοτήτων. Παρά το γεγονό ότι υπήρχε χειροθέτηση από κάποιε ομάδε ε, τα τελευταία χρόνια, δεν θα έλεγα ότι όλοι υποστηρίζουν πλέον τόσο αναφαντών τον κύριο Μοράλε. Θα ήταν θεκτικό τα επόμενα χρόνια να δούμε ελεύθερε εκλογέ με διαφορετικού υποψηφίου χωρί ε, παρεμβάσει. Ξεκινά λοιπόν σήμερα και σε υψηλό επίπεδο διάλογο στη Λαπά. Η βλέπουμε το ζήτημα της συνεργασίας με τη Βολιβία και στο γενικότερο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας ε, είναι ε, προσωρινό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτή τη στιγμή η Βολιβία. Όμως δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι υπερψηφίζει ψηφίσματα και παίρνει τις θέσεις α, χωρών που δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς φιλικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ακολουθεί τη δική μας γραμμή. Το ανέφερε και ο κύριος Τσέλαρ ε, Κοιτούμε γενικότερα λοιπόν το ζήτημα της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, αλλά επίσης και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Σε αυτούς τους τομείς θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος με τη Βολιβία. Και επίσης θα θέλαμε να δούμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών της κοινωνίας στα, στα κοινά, στα διάφορα επίπεδα της πολιτικής στη χώρα. Ε, επαναλαμβάνω λοιπόν ότι συμφωνούμε με πολλές από τις παρατηρήσεις που, γίνω, που σε σχέση με τη συνεργασία αλλά συμφωνούμε επίσης και στις παρατηρήσεις που, γίνονται, που έγιναν από τον κύριο Τσέλερ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. θεωρούμε ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία, αλλά ακόμα μπορεί να γίνουν πολλά και να ε, σημειωθεί πολύ μεγαλύτερη πρόεδρο σε αυτή τη χώρα. Σα ευχαριστούμε. Θα ήθελα να προσθέσει κάτι η Δεύκο και μετά θα δώσω το λόγο στον άλλο συνάδελφο, του κ. Τεμέρο, Αγουστίν. Μετά, μετά τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, Αγουστίν, μπορείτε να. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ για την έκθεση αυτή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά θετικά πορίσματα στην αποστολή αυτή και όπως υπόθηκε στηρίζουμε τις αρχές της Βολιβίας καθώς επίσης και τη συμβολή του Εύω Μοράλες ο οποίο συμβάλλει και αυτό σε συνεργασία μεταξύ Βολιβία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τη συνεργασία, η Βολιβία είναι μια πολύ σημαντική χώρα γιατί όχι μόνο λαμβάνει σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της Λατινικής Αμερικής, αλλά είναι και ο μεγαλύτερος, αν θέλετε, δικαιούχος της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να επικεντρωθούμε σε όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η αποστολή αυτή. Εμείς ε, προσπαθούμε να, επιβάλλουμε να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου η δική μας η παρέμβαση να είναι στο δυνατόν πιο αποδοτική και αποτελεσματική, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης αλλά και σε άλλους τομείς. Λαμβάνουμε υπόψη τα πορίσματα της αποστολής αυτής, συμφωνούμε τα συμπεράσματα της έκθεσης και θεωρούμε ότι όντως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ε, σημασία στο περιβάλλον, στην ε, καλύτερη διαχείριση των υδάτων, καθώ επίση και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματο. Τι επόμενε εβδομάδε θα υποβάλουμε δύο νέα προγράμματα στον τομέα τη δικαιοσύνη, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε στο μέλλον μια πιο σημαντική παρέμβαση στον τομέα αυτή και μια ακόμα σημαντική παρέμβαση θέλουμε να έχουμε όσον αφορά την εξυγίανση των υδάτων στι πόλει και στην Ήπεθρο. Ελπίζω ότι τα δύο αυτά προγράμματα θα εγκριθούν πριν το τέλο του έτου. Σα ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο Αγουστίν Διάς Δεμέρα τώρα έχει το λόγο, παρακαλώ. We heard Ακούσαμε τους άλλους δύο συναδέλφους που ήταν μαζί σας στην αποστολή. Ναι, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, και να ζητήσω συγγνώμη και από εσά και από όλου του συναδέλφου που καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να ψηφίσω στην ε, Επιτροπή Λίμπε. Ποια είναι η εντύπωση που αποκόμισα από την αποστολή μας. Θα έλεγα ότι ήταν θετική, πολύ θετική για τον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοι, η κυρία Θεοχάρους και ο κύριος Φρουντζούλητσα ε, λειτουργήσαν και επίσης ε, πολύ θετική για την αποτελεσματικότητα της γραμματείας και των συναδέλφων που μας υποστήριξαν. Τους ευχαριστώ πολύ. Συζητούμε για, συζητήσαμε για τρία θέματα, την δικαιοσύνη και την ε, διαφθορά, του, τα ναρκωτικά και το, τα ύδατα, το νερό. Πρέπει να πω ότι σέβομαι την κυβέρνηση της Βουλιβίας και τον πρόεδρο τον κύριο Μοράλες παρά το γεγονός ότι έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Είχα, μας ε, φιλοξένησαν και μας υποδέχθηκαν ε, εξαιρετικό τρόπο. Είχαμε συναντήσει σε υψηλότατο επίπεδο με τέσσερις υπουργούς και έναν υφυπουργό και πολλούς άλλους. Και φαντάζομαι ότι ήδη θα θα διαβάσατε την αναλυτικότατη έκθεση και θα το συζητήσατε. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η καταπολέμηση των παράνομων καλλιεργειών κόκας και η κατάστασή τους με νόμιμες καλλιέργειες. Ε, ο κύριος Μοράλες που προσπαθεί να αξιοποιήσει την ζώνη του τροπικού που βρίσκεται στην Βολιβία για να δώσει εναλλακτικέ και να να δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές καλλιέργειε για να αντικαταστήσουν το, την κόκα. Ε, σπυριδοειδή, ε, μάγκο ε, και... κάποια είδη, κάποια, κάποια, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την διατροφή των αυτοχθόνων αλλά επίσης και για εξαγωγές. Είχαμε επίση συναντήσει σε υψηλό επίπεδο ε, με εκπροσώπου γυναικών από την κοινωνία των πολιτών και μπορεί κανεί να διαπιστώσει ότι γίνεται πολύ καλή και αποτελεσματική χρήση των ε, χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνουν για την ενδυνάμωση των γυναικών, για την εκπαίδευση ε, ε, γυναικών ηγετών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, για την εκπαίδευση των ανθρώπων στις σωστές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Ε, και θα έλεγα και, επίσης για να μπορέσουν οι γυναίκες να αυτονομηθούν και να χειραφητηθούν και να είναι ε, ανεξάρτητες μέσω της δουλειάς τους. Θα έλεγα ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικό και στην προηγούμενη μας... πάλι, ε, στην, στην ε, συνάντηση που είχαμε με τους ειδικού. Με είχα την τιμή να συναντήσω και εκπροσώπους ε, του, στρα, στρατού της Βολιβίας με τους οποίους συζητήσαμε το ζήτημα της, της ε, συνεργασίας για την καταπολέμηση του εμπορίου των ναρκωτικών. Ε, θα έλεγα ότι είναι γενικές γραμμές πολύ επιτυχημένη η αποστολή μας και θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους για αυτήν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα είπατε. Νομίζω ότι μα ε, μας έγινε μια διεξοδική παρουσίαση πλέον της αποστολής αυτής. Το επόμενο κοινοβούλιο βέβαια θα πρέπει να δώσει συνέχεια σε συνεργασία αυτή με τη Βολιβία. Μας απομένουν τέσσερις μήνες. Παρ' όλα αυτά γίνονται κάποιες συστάσεις στην έκθεση οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, το προσωπικό που συμμετείχε στη διοργάνωση αυτής της αποστολής, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, καθώς επίσης και τους εργοζομένους Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιπροσωπεία που έχουμε στην ε, Βολιβία. Περνάμε στο σημείο 19 της της διάταξης, όπου ε, συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η Ελένη Θεοχάρους, Συμφωνία Αλλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Δημοκρατίας της Ακτής του Λεφαντοστού και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος. Εδώ πέρα έχουμε τόσο τη γνωμοδότηση αυτή καθεαυτή, όσο και τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Η Επιτροπή Αλίας μας ε, ενημέρωσε ότι θα ψηφίσουν τον Ιανουάριο για τη νέα αυτή συμφωνία αλληλευτική σύμπραξη. Γι' αυτό το λόγο πιέζει αρκετά ο χρόνο. Πρέπει σήμερα να γίνεται αλλαγή απόψεων και προβλέπεται στι 10 ή 13 Δεκεμβρίου μια έκτατη συνεδρία τη Επιτροπή μα στο Στρασβούργο. Να ξαναδώσω πάλι το λόγο στην Ελένη Θεοχάρου για να μα ενημερώσει για το ζήτημα αυτό. Ελένη, έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω τα σχετικά με το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο θα συναυθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού και θα πρέπει να συνάδει πλέον με τον κανονισμό της νέας κοινή ελευτικής πολιτικής, που ε, εστιάζει κυρίως στην χρηστή διακυβέρνηση και την βιώσιμη αλία και προβλέπει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια ανάμεσα στην κοινή ελευτική πολιτική και τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασία και καλύπτει το πρωτόκολλο αυτό μια εξαιτή περίοδο για μεγαλύτερη σταθερότητα. Η πρόσβαση των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στους ελευτικούς σπόρους, τους οποίους η ακτή του ελεφαντοστού δεν διαθέτει την ικανότητα να εκμεταλλευτεί. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στα πλεονάσματα των πόρων και θα πρέπει εδώ πέρα να ακολουθήσουμε και τα όσα λέει η, η κάρτα προβλέπεται εδώ πέρα ένα συνελικό ποσό 5.500 τόνων, το οποίο είναι χαμηλότερο από αυτό το οποίο προβλεπόταν στο παρελθόν. Βλέπουμε παρόλα αυτά όμως ότι δίνεται δυνατότητα για συγκεκριμένες ζώνες αλίευσης για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ πέρα μπορούμε ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε και τις άλλες συμφωνίες που έχουμε συνάψει με άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια, ένα ευρύ δίκτυο αλίευσης στο οποίο μπορεί να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ζητώ συγγνώμη αυτή τη στιγμή, δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω αυτά τα οποία έχω μπροστά μου γιατί είναι αρκετά μικρά τα γράμματα. Πάντως, η χρηματοδότηση προβλέπεται εδώ πέρα στο νέο αυτό πρωτόκολλο 628.000 ετησίως ευρώ αποτελούν μια αύξηση σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα δύο πρώτα χρόνια το σύνολο αυτό ουσιαστικά θα είναι 330.000 το πρώτο σκέλος για την πρόσβαση στην ελευτική ζώνη της ακτής του Λεφαντοστού, ενώ τα υπόλοιπα 352.000 ευρώ θα πάνε στον ειδικό σκοπό της στήριξης εφαρμογής ελευτικής πολιτικής στην ακτή του Λεφαντοστού. Τώρα για την υπόλοιπη περίοδο το ποσό θα είναι 275.000 ευρώ και 407.000 ευρώ αντίστοιχα. Πρόκειται για μια σημαντική και πρόσδεκτη αύξηση του τομεακού προπολογισμού η οποία βασίζεται στην βιώσιμη αλίευση και στην πιο υπεύθυνη αλία και έχει ως στόχο να υποστηρίξει την αλία μικρής κλίμακας, τη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για τα ίχθη αποθέματα, τη στήριξη της γαλάζιας οικονομίας και την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Θεωρώ ότι το πρωτόκολλο αυτό θα προαγάγει την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των ελευτικών πόρων στην ακτή του ελεφαντοστού προ το συμφέρον και των δύο μερών και ότι ω εκ τούτου συνάδει με του στόχου των συμφωνιών βιώσιμη Αλληλεία και τη αναπτυξιακή συνεργασία. Για του λόγου αυτού, προτείνω να εγκριθεί αυτό το πρωτόκολλο. Αυτό το οποίο προτείνουμε λοιπόν σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας Επιτροπής Αλίας είναι να επικεντρωθούμε κυρίως στην ανάπτυξη της παραδοσιακής αλίας και της αλίας μικρής κλίμακας και να δημιουργηθούν οι απαραίτητε συμφωνίε εταιρική σχέση στον τομέα αυτό. Να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο την συμμετοχή των γυναικών, να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση του τομέα τη αλίας, για να καταφέρουμε να αποφύγουμε την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία και θέλουμε επίση να έχουμε και την απαραίτητη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση τη τομεακή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πρωτοκόλου αυτού, προκειμένου να παρακολουθούνται και να βελτιώνται τα ποσοστά απορρόφηση και να διασφαλίζονται έτσι ότι η συμφωνία αποφέρει απτά αποτελέσματα και στήριξη τη τοπική αλληλεία και του τοπικού πληθυσμού γενικότερα. Σα ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ποιοι άλλοι θέλουν να πάρουν το λόγο, κύριο Πόγκα. Καλώ ήρθατε πάλι στην Επιτροπή μα. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο, την κυρία Θεοχάρους, για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης και θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή της. Πραγματικά θα πρέπει να εγκρίνουμε το πρωτόκολλο αυτό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να στηρίξουμε τις προσπάθειες της ακτής του ελεφαντοστού προκειμένου να έχει και αυτή μία αλληλεία η οποία να είναι βιώσιμη. Αυτό είναι προς το κοινό μας συμφέρον θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες ε, στο ψήφισμα αυτό, λέγοντας ουσιαστικά ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε την ακτή του Λεφαντοστού να καταπολεμήσει την παράνομη και λαθρέα αλία, προκειμένου να αυξηθεί επίσης και η διαφάνεια εφαρμογή του πρωτοκόλου αυτού και προκειμένου να έχουμε και μια ετήσια έκθεση για την υλοποίηση του πρωτοκόλου αυτού, έκθεση η οποία θα πρέπει να διαβιβάζεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σα ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε ο κύριος Κορνιέ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως θα πρέπει να συνδυάσουμε την γνωμοδότηση αυτή με κάποιους άλλους τομείς. Ξέρετε ότι στα πλαίσια της γαλάζιας ανάπτυξης η αλληλεία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα δίπλα σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός. Όπως είπε και η συνάδελφος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη συμφωνία αυτή με την ακτή του Εθαντοστού, αλλά η συμφωνία αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί και με τις αλλιευτικές συμφωνίες που έχουμε με τις υπόλοιπε περιοχές της Αφρικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ο, απόλυτο, ο απαραίτητος συντονισμός και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πέρα από την συμφωνία των πράξεων αυτών χρηματοδότησης, όπως είπε και ο κύριος Πονκά, θα πρέπει να έχουμε και μια ετήσια έκθεση όχι αναγκαστικά αναχώρα, αλλά τουλάχιστον ανααλλιευτική ζώνη, η οποία να φτάνει και σε εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ ότι όλοι οι συνυπογράφοντε το πρωτόκολλο αυτό όντω τηρούν του κανόνε που περιέχονται σε αυτό το πρωτόκολλο. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να το διασφαλίσουμε και θα καταθέσω μια σχετική τροπολογία. Πολύ ωραία. Αυτό θα έλεγα και εγώ, λέει η Πρόεδρο, ότι εφόσον θέλετε να περάσουν τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να καταθέσετε και σχετικέ τροπολογίε. Ο κύριο Τζέλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε μια στον χρόνο του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά αυτή την εταιρική σχέση. Μέχρι σήμερα δεν μου είναι ξεκάθαρο πώς αυτά τα πλεονάσματα ε, υπολογίζονται. Υπάρχουν ε, μέθοδοι επιτήρησης πιο πολλές από αυτές τις χώρες. Όταν υπάρχουν και γνωρίζουμε ότι ο τόνος είναι ένα ψάρι και όχι μόνο τόνος, αλλά και άλλα ψάρια που έχει μια μεγάλη περιοχή που είναι πρακτικό σε, μια μεγάλη περιοχή, ένα, σε μεγάλο ζωτικό χώρο. Όμως, ε, επιμένουμε να ενισχυθεί η τοπική αλία. Είμαστε στην Ελλάδα φέτος για να δούμε και τη βιομηχανία την αλληλευτική. Ήταν οι συνθήκε εργασία, για πιστού από ένα εκατομμύριο μετανάστες εργαζόμενου στην, στον τομέα της αλληλείας, αλλά αυτό που μας είπαν εκεί οι αρμόδιοι ήταν ότι δεν θα υπάρχει τόνος στο μέλλον, ότι υπάρχει, πουλάνε κονσέρβες τόνοι, οι δεν έχουν μέσα τόνο, αλλά μπορεί το ένα παρόμοιο ψάρι με τον τόνο. Τώρα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αλληλευτικά σκάφη και τα ισπανικά έμαθα από την Επιτροπή ότι πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι στην Ιαπωνέζικη αγορά, γιατί εκεί τα στάνταρ της ποιότητας είναι πολύ πιο υψηλά. Thank you very much. I think there's somebody from DJ Mare here. Σα ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιο εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας. Μάρε. Ναι. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Είχα μια εμπειρία από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχαμε συζητήσει πολλές φορές τα ζητήματα αυτών των συμφανιών αλίας και το τι αποτελέσματα επιπτώσεις μπορεί να έχουν όχι μόνο για την πρόσβαση στην αγορά αλλά και για το ζήτημα της βιωσιμότητας. Θέλετε να μας δώσετε περισσότερε πληροφορίε να έχουν και οι συνάδελφοι μια καλύτερη εικόνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Σα ευχαριστώ για τι παρατηρήσει σα για αυτήν τη συμφωνία αλίας και για το γενικότερο πλαίσιο των συμφωνιών αλίας που πρέπει να προωθούν τη βιωσιμότητα και με τις οποίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα συμφωνιών με χώρες της Αφρικής και του Ειρηνικού. Πράγματι, εδώ, μιλώντας για την ακτή του ελεφαντοστού, μιλούμε για αλία τόνου, κυρίως από γαλλικά και ισπανικά αλλιευτικά, με μεγάλες ποσότητες ε, τροπικού τόνου. Δεν μιλάμε για τον κόκκινο τόνο εδώ. Που πράγματι πολλούνται κυρίως στην ε, η Ιαπωνική αγορά ο κόκκινος τόνος, ενώ ο τροπικός τόνος κυρίως πηγαίνει προς την Γκάνα ε, ή προς τις Σίγελες. Επομένως, είτε επεξεργασμένα, ε, ε, μετά από επεξεργασία, μεταποίηση, γίνεται η εξαγωγή, είτε γίνεται η συσκευασία σε κονσέρβες στην ακτή Λεφαντοστού και στην ε, Γκάνα. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε επιπλέον ότι είναι σημαντική η συμφωνία με την ακτή Λεφαντοστού γιατί υπάρχει και αυτή η βιομηχανία της ε, ε, επεξεργασίας του ψαριού επιτόπου και έμεσα βοηθείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και τα ελευτικά φέρουν σημαίες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της βιώσιμης αλίας του τροπικού τόνου ε, το αντιμετωπίζουμε στο περιφερειακό επίπεδο, γιατί όπως σωστά είπατε δεν περιορίζεται το απόθεμα μόνο στην, σακτές μιας χώρας, αλλά σε μια ολόκληρη περιοχή Γι' αυτό υπάρχει αυτή η περιφερειακή συνεργασία, για να υπάρχει μια γενικότερη ε, συνεργασία στην περιοχή του Ατλαντικού. Υπάρχει μια διεθνή Επιτροπή για τον τόνο του Ατλαντικού, η ΣΥΚΤΑ, η οποία συναντάται τεκτικά, εξετάζεται επιστημονικά δεδομένα και επί τη βάση αυτών κάνει προτάσεις για το ποιος, ποια πρέπει να είναι η ποσόστοση. Η ποσόστοση εφαρμόζεται και στα ευρωπαϊκά ε, ε, ε, σκάφη, τα ευρωπαϊκά σκάφη βεβαίω αξιοποιούν την ποσόστοση που αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την ποσόστοση που αντιστοιχεί σε αυτέ τι χώρε. Δεν βρισκόμαστε στα χωρικά υδατά. Η αλληλεία αυτή γίνεται αρκετά μακριά στα, στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν επίσης και μέτρα για την υποστήριξη των μικρών αλλιέων ε, που έχουμε διατυπώσει σε συνεργασία με την ε, χώρα εταίρο ε, ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες που μπορεί να έχουν αυτά τα μικρά αλλιευτικά και οι, οι, Τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε και άλλες συναντήσεις με τους εκπροσώπους της ακτή ελεφαντοστού έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα που και εσεί αναφέρετε, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της παρακολούθησης, ε, της ηχνηλασιμότητα. Ε, και επίσης για το ζήτημα των μικρών αλλιών. Θα έλεγα ότι για το ζήτημα των μικρών αλλιών, ιδιαίτερα το εκτήλεφαντος του, είναι χώρα υπόδειγμα. Γιατί υποστηρίζουμε και μέτρα έτσι ώστε να μπορούν να, να, ε, πολλούνται και τα παράπλευρα αλλιεύματα, άλλα ψάρια που πιάνει κανείς ενώ δεν ήταν αυτό που στόχευε, και να γίνεται απόθεση αυτών των παράπλευρων αλληλευμάτων όταν φτάνει το πλοίο στην ακτή ελεφαντοστού για να μπορούν μετά αυτά να απολυθούν και να αξιοποιηθούν εμπορικά και, ε, και τα λοιπά και για μεταποιημένα τρόφιμα στην ακτή ελεφαντοστού. Θα έλεγα ότι αυτό είναι μια καλή πρακτική, ένα καλό παράδειγμα γιατί βοηθάει και την τοπική οικονομία ε, με έναν επιπλέον τρόπο. Όσον αφορά την παρακολούθηση, η χώρα αυτή ε, θα έχει τη δυνατότητα με βάση τη συμφωνία να κάνει ε, αναγνωριστικές επισκέψεις ε, είτε σε, σε, σε αλλιευτικά είτε με, με, με σημαία Ένωσης και παράλληλα ο, ο Ευρωπαϊκός Στόλος θα έχει ένα δικό του πρόγραμμα εθελοντικό για τους ελέγχους, ε, την παρακολούθηση έτσι ώστε αυτή να είναι εξαντλητική. Ιδίω για τα μεγάλα αλληλευτικά. Το Ιεκτή ελεφαντοστού λοιπόν θα συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα Ελέγχω. Όσον αφορά το reporting. Έχουμε μια μεικτή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν όλες, όλοι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή της συμφωνίας και η οποία θα καταλήγει σε μια έκθεση, θα συνυπογράφεται από τα δύο μέρη και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή θα αποστέλλεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα μας δίνει στοιχεία και όσον αφορά τους προϋποθέσεις που τίθενται για την πρόσβαση του στόλου μας στις περιοχές αυτές, αλλά και επίσης για άλλα αριθμιστικά στοιχεία ε, παρακολούθησης. Θα υπάρχει επίσης και σε αιτήσια βάση μια ε, έκθεση για την υλοποίηση της συμφωνίας. Επομένως θα έλεγα ότι το ζήτημα της διαφάνειας και της ενημέρωσης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου έχει καλυφθεί επαρκώς. Τώρα, το πώς συνδέονται αυτή η πολιτική με την πολιτική ανάπτυξη, νομίζω θα το αναπτύξει περισσότερο η συνάδελφος, θα έλεγα πάντως ότι υπάρχει και προσπαθούμε να χτίσουμε και σε ένα περιφερειακό επίπεδο αυτό το, το πρόγραμμα ελέγχων. Σας ευχαριστώ. Ε, νομίζω πω το Μαριάν ακούσαμε από το Μάρι. Για το πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση, είχαμε καλά παραδείγματα από στην Κάνα, όπου δημιουργήθηκαν θέσει εργασία και δημιουργήθηκαν και επαγγελματα στον τομέα τη μεταποίηση. Ελένη, θα ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο. Λοιπόν, την 5η 10 η ώρα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 13 Δεκεμβρίου, μάλλον, Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο ε, Στρασβούργο. Θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε άργιε συνεδριάσει όπω την προηγούμενη φορά που είχαμε 9 ώρα συνεδρία στο Στρασβούργο. Θα δούμε πώ το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο σημείο 21 που είναι η κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού. Προχωράμε στο σημείο 21 την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού το 2018. Θα μιλήσουμε για την έκθεση, για την έκθεση του 2018 για την κατάσταση του πληθυσμού που εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό. Ε, ο τίτλος είναι «Η δύναμη της επιλογής, αναπαραγωγικά δικαιώματα και δημογραφική μετάβαση». Θα... Η κυρία Σίσκετ Στένεκε θα μας μιλήσει, που είναι η πυρογνώμονας Μίλησαμε σε μια συνεδρίαση για τη στάση της γονιμότητας η οποία ε, έχει πέσει τα τελευταία 100 χρόνια μας υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών. Συναντήθηκα με υπουργό από τον Ήγηρα όπου ε, έχουμε 7 παιδιά ένα οικογένεια. Ενώ στις δικές μας χώρες έχουν πέσει δραματικά τα ποσοστά της γονιμότητας στην Ιαπωνία έχουν πρόβλημα και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Για μένα προσωπικά ένα θέμα που μας ενδιαφέρει είναι η επιλογή των γυναικών στο θέμα της γονιμότητας. Κάτι που έχουμε την τύχη στις χώρες μας να το έχουμε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Τένικη για 10 λεπτά και μετά θα δώσω το λόγο ε, στα μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ε, την έκθεση τη φετινή για την κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχει να κάνει με τις τάσεις γονιμότητας στον κόσμο, αλλά και με την ε, ύπαρξη επιλογής, την έλλειψή τη για τις γυναίκες, τα ζευγάρια, αλλά και για τις χώρες και τις προοπτικές για εξέλιξη όταν ε, ετοιμάσαμε την εκθέση, πήραμε συνέντευξη από άτομα από όλο τον κόσμο. Πρωτού σα δώσουμε το γενικότερο περιεχόμενο, θα ξενικήσω με μικρά βίντεο που δείχνουν τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Βλέπουμε τη Σάρο στο Ναϊρόμπι που ζει με την οικογένειά της. Is eight years old. My second is a girl. She will be two years old in June. We don't plan to have more children because of the situation in Kenya. There is no money. So the two will be fit for us to get a from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 try to support my husband. Like many Kenyans today, όπως πολλοί Κενιάτες, η Σάρο και ο σύζυγός της προτιμούν να έχουν λιγότερα παιδιά για να μπορούν να φροντίσουν καλύτερα αυτά που έχουν. Θα ήθελα να δείξω ακόμα ένα βίντεο, αλλά θα το παραλείψουμε. Η πρόεδρος επιμένει να το δείξει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 11 δείχνει τη σημασία των δημόσιων πολιτικών που βοηθούν στην Σουηδία, παραδείγματος χάρη, ε, με την άδεια να για τους πατέρες και δίνουν τη δυνατότητα στα, ε, στις οικογένειες να αποκτήσουν τα παιδιά που επιθυμούν και παράλληλα να έχουν την καριέρα τους. Θα ήθελα να αναφερθώ τι εννοούμε με την έννοια της επιλογής. Έχει να κάνει με το να έχει κάποιος τα μέσα και την δυνατότητα να ε, αποφασίζει μόνος του πότε και πόσα παιδιά θα κάνει και πόσο επηρεάζει και τους άλλους. Αναφερόμαστε και στα παραγωγικά δικαιώματα και τους παράγοντες που εμποδίζουν ή ε, καθιστούν δυνατή την ε, λήψη τέτοιων αποφάσεων Φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια είναι η ισότητα μεταξύ των φύλων, όπου οι γυναίκες έχουν δυνατότητα να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Είναι πολύ σχετικό και με την εβδομάδα σχετικά με την εβδομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων το 1910. Ε, σύνοδο αυτή λοιπόν αποφάσισαν ότι είναι σημαντικό η κάθε οικογένεια να αποφασίζει μόνη της τον αριθμό των παιδιών. Ε, τα άτομα έχουν αναπαγωγικά δικαιώματα και οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να εμποδίσουν ή να καθυστερούν τις εγκυμοσύνες. Ε, στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, 671 εκατομμύρια γυναίκες έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, αλλά υπάρχουν 214 εκατομμύρια γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο που ε, διατρέχουν κίνδυνο να μείνουν ε, έγκυες χωρίς τη θέλησή τους. Ε, σε πολλές επίσης χώρες οι γυναίκες γίνουν περισσότερα παιδιά από όσα θα ήθελαν. Στις πιο αναπτυγμένες χώρες είναι περιορισμένη και εκεί η επιλογή. Σε χώρες χαμηλής γεγονιμότητας, μπορεί να, ε, να εμποδίζεται αυτή η επιλογή εξαιτία του υψηλού κόστους ε, για τη φροντίδα των παιδιών και γι' αυτό πολλέ ε, γυναίκε έχουν λιγότερα παιδιά από όσα θα ήθελα. Ε, το κατά πόσο έχουν την επιλογή αυτή οι γυναίκε θα επηρεάσει τι ε, τάσει τη γονιμότητας μακροπρόθεσμα. Υπήρχε ένα ποσοστό γονιμότητας μέχρι πρόσφατα, ένα υψηλό ποσοστό γονιμότητας, έξι γένες ανά γυναίκα. αλλά τα ζευγάρια ήθελαν και κατάφεραν να έχουν μικρότερες οικογένειες προτού ε, υπάρξουν διαθέσιμοι μέθοδοι αντισύλληψης και παρά την πίεση από την κοινωνία και από τη θρησκεία. Μόλις το κατάλαβαν αυτό στην Ευρώπη άρχισαν να επιλέγουν τις μικρότερες οικογένειες και καθώς τα ζευγάρια σε άλλα μέρη του ε, κόσμου απέκτησαν και εκεί την ε, δυνατότητα επέλεξαν επίσης να έχουν μικρότερες οικογένειες. Το βλέπουμε αυτό στο επόμενο σχέδιο που βλέπετε την ε, δημογραφική μετάβαση. Το 1800 ε, ο αριθμός παιδιών ένα γυναίκα ήταν γύρω στα 6. Σε κάποια μέρη υψηλότερη ή χαμηλότερα, αλλά ήταν υψηλό το ποσοστό όπως και να έχει παντρεύονταν νωρί, δεν είχαν κατανόηση για, για την έννοια τη σύλληψη, ε, η παιδική θνησιμότητα ήταν ψηλή, το προσδόκιμο τη ζωή χαμηλό και το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα ήταν υπέρ των μεγάλων, ε, ε, μεγάλων οικογενειών. Είχαμε όμω μια αλλαγή. Από τα έξι παιδιά πέρασαμε σε λιγότερα από δύο παιδιά μέσα σε 100 χρόνια. Ε, το, δεδομένο, το ζητούμενο ήταν να κρατήσουμε το επίπεδο του πληθυσμού στο ίδιο επίπεδο. Επίσης είχαμε πτώση και στι Ηνωμένε Πολιτεία και στις άλλες χώρες, ε, τι αγγλόφωνε χώρε όπως η Αυστραλία. Έχουμε μια καθυστέρηση στην ε, Ευρώπη. Βλέπετε ε, την ανωδική καμπύλη σε εκείνο το σημείο. Ήταν μια νέα τάση τότε με τον baby boom. Επίσης έχουμε και την κόκκινη ε, καμπύλη που αντιστοιχεί στην Ασία. Ξεκίνησε αργά αυτή η τάση στην Ασία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν πολύ γρήγορη. Αυτό που χρειάστηκε 200 χρόνια να συμβεί στην Ευρώπη συνέβη σε μισό αιώνα στην ε, Ασία. έχουμε και την Αφρική, την Black καμπύλη. Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε και εκεί μία πτώση, όχι όμω όσο γρήγορα όσο σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν επίσης ε, ε, βλέπουμε ότι έχουμε πιο γρήγορη μείωση της γονιμότητας στην Αφρική σε κάποιες χώρες είναι κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης του πληθυσμού, κάτι που έχει συμβεί στην Νότια Ευρώπη και στην Ανατολική Ευρώπη, όπως και στην ε, Ιαπωνία, στην Κορέα και στην Αυστραλία. Βλέπουμε ότι η... τα ποσοστά γονιμότητας είναι διαφορετημένα όσο ποτέ. Σε κάποιες χώρες έχουμε 7 γυναίκες 7 παιδιά, συγγνώμη, ανά γυναίκα, όπω είναι στην Νιγηρία και σε άλλε χώρε τη Ποσαχάρη Αφρική, όπου είναι πολύ υψηλό το ποσοστό, ενώ σε άλλε χώρε τα ποσοστά γονιμότητα αγγίζουν το ένα παιδί ανά γυναίκα. Αναφέρομαι στην Ταϊβάν. Ανεξάρτητα από το αν είναι υψηλή ή χαμηλή γονιμότητα, ε, αποτελεί πρόκληση για τις οικονομίες, τις, ε, τους θεσμούς και τις ε, πρακτικές και το μέλλον μιας χώρας οι χώρε υψηλή γονιμότητας ε, αγωνίζονται για να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στον ε, ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό. Στις ε, χώρε χαμηλή γονιμότητας δυσκολεύονται να διατηρήσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και να έχουν το παρέτητο εργατικό δυναμικό για τις οικονομίες τους. Εμπλέκονται φυσικά εδώ και τα δικαιώματα και οι επιλογέ. Πολλέ χώρες ε, επέλεξαν ε, να περιορίσουν τις επιλογέ και να παραβιάσουν τα δικαιώματα των γυναικών. Η κατάσταση του παγκόσμιου πληθυσμού ζητάει να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι επιλογέ. Αυτό θα ήταν το σωστό και για τα άτομα και για τα ζευγάρια αλλά και για τις κοινωνίες στο σύνολό τους αν δούμε την ε, δημογραφική μετάβαση, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η επιλογή μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί και ραγδαία να βελτιώσει την ε, ευημερία των γυναικών και να επιταχύνει την παγκόσμια ανάπτυξη. Η έκδοση αυτής της ε, έκθεσης είναι μια νέα προσπάθεια ε, του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Παγκόσμιο Πληθυσμό να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τις επιλογές για όλους. Στον επόμενο χρόνο θα έχουμε μια ε, ε, διεθνή σύνοδο για τον πληθυσμό και την εξέλιξη. το ICPD συγκεκριμένα, το οποίο ήταν εξαιρετικό στο να αναγνωρίσει τη σημασία της αναπαραγωγικής υγείας των δικαιωμάτων. Έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδο, όμω έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μα. Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ακόμα 99 εκατομμύρια ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε, γιατί οι γυναίκε δεν έχουν επιλογέ αντισύλληψη. Κάθε χρόνο πάνω από 300.000 γυναίκε πεθαίνουν κατά τη διάρκεια τη ε, εγκυμοσύνη ή του τοκετού, επειδή δεν έχουν επιλογέ ε, όσον αφορά ε, την η υγειονομική περίθαλψη. Κάθε μέρα δεκάδες ε, χιλιάδες υποχρεούνται να παντρευτούν και γίνονται μητέρες ήδη στην εφηβεία, χωρίς να έχουν επιλογή. Πρέπει να επεκτείνουμε την επιλογή σε όλους αυτούς που έχουν μείνει πίσω, έτσι ώστε ως το 2030 ο χρόνος που είχε οριστεί για την επίτευξη των των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων θα πρέπει να έχουμε ε, τη δυνατότητα να έχουν όλοι πρόσβαση σε αντισύλληψη και να μπορούν να αποφυγούν τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Χρειάζεται παγκόσμια συνεργασία για να ενισχύσουμε ε, την, ε, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών Φυσικά οι ευρωβουλευτές έχουν ε, να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να υψώσουμε λοιπόν τη φωνή μας, να ενημερώσουμε σε σχέση με την... Ε, να σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, ενημέρωση σωστή και όλα αυτά να προβληθούν και στο πολιετές φυσικά ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όντω, οι διαφάνειε που μα δείξατε καταδεικνύουν πάρα πολύ καλά πώ έχουν τα πράγματα. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια εννιά παιδιών. Οι γονεί μου ήταν καθολικοί και την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 60 και του 70, ήταν πολύ μεγάλες οι οικογένειε, πολύ ήταν οι πολίτεκνοι, ενώ τώρα είναι κάτι το οποίο σπανίζει. Η έκθεση πάντω είναι πάρα πολύ καλή αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ την ανέτρεξα γρήγορα και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν προσωπικές μαρτυρίες από διάφορες γυναίκες. Μια γυναίκα από τη Βραζιλία 87 ετών λέει ότι απέκτησε 22 παιδιά ή τουλάχιστον είχε την εμπειρία 22 γεννήσεων. Όταν αναφερόμαστε εδώ πέρα σε φαντάζομαι ότι αναφερόμαστε όχι σε παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, όχι σε εγκυμοσύνες. Οι γυναίκε αυτέ τι οποίε αναφέρατε στην εκκλησία προφανώς είχαν πολύ περισσότερε εγκυμοσύνες και χρειάστηκε κάποια στιγμή ενδεχομένω να αποβάλουν κτλ. Αναφερθήκατε στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αναφερθήκατε στα νέα μέσα τα οποία έχουμε. Έχουμε τον συνεισηγητή μα εδώ πέρα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Επομένω άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε για την επιλογή και κυρίω για την επιλογή οικογενειακού προγραμματισμού δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι που θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Σάρλ, ξέρω ότι έχει ολοκληρώσει την εκθεσή σου, επομένω ε, μπορεί να μα μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον ε, ζήτημα το οποίο προκύπτει και το οποίο θα μπορούσαμε να θέσουμε ως ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προς το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό είναι ότι ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση της εργασίας για το NDCI και το έγγραφο αυτό τώρα βρίσκεται στη φάση της μετάφρασης, θα κοινοποιηθεί, θα δημοσιευθεί σε μερικές ημέρες. Διερωτώ με όμως ε, από ποια πλευρά εμείς μπορούμε να επέμβουμε, να βαρύνουμε λίγο περισσότερο στις επιλογές που γίνονται. Χρησιμοποιήστε και εσείς τον όρο επιλογή. Επιλογή προγραμματισμού, οικογενειακού προγραμματισμού. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ζητήσαμε μια ευρύτερη συμμετοχή στο πλαίσιο της εργασίας αυτής που κάναμε, οι τέσσερις συνεισηγητές. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε είναι να μπορούμε να βαρύνουμε περισσότερο και να πειράσουμε τις κύριες προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επίσημη οικονομική βοήθεια, την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, θέλουμε να δούμε αν στα πλαίσια του μελλοντικού προγραμματισμού θα υπάρχει μία συγκεκριμένη πλέον στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την λεγόμενη διαχείριση των δημοκρατικών τάσεων. Βλέπουμε ότι στην περιοχή του Σαχέλ οι δημογραφικές τάσεις είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονες, ενώ από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες προσπαθούν να ρυθμίσουν τις γεννήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει μέσω των κατεξοδότηση πράξεων να έχουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες και ως Ευρωβουλευτές αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορούμε εμεί ε, να συμβάλλουμε, να επηρεάσουμε τα πράγματα. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον. Ελπίζω να καταφέρουμε να αυξήσουμε τι αρμοδιότητε μα. Το σημαντικό είναι το νέο αυτό εργαλείο, το νέο μέσο να τεθεί σε ισχύ και αν ε, διατηρηθεί με τη μορφή που το υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον τρόπο που τροποποιήθηκε τελικά από τους τέσσερις ενησυγητές, θα θέλαμε να γνωρίζουμε συγκεκριμένα την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής Παρευρίσκεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι έχει συμβάλει πολύ στο μέσο αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και μια στρατηγική εταιρική σχέση, προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμεί στην εξέβρεση λύσεων. Αν πάρετε μια χώρα σαν το Κονγκό, θα δείτε ότι στην Κινσάσα, την πρωτεύουσα, έχουμε μια αύξηση ετήσια 300.000 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν και τα απαραίτητα εκπαιδευτικά ιδρύματα που να μπορούν να απορροφήσουν όλα αυτά τα παιδιά. Ποιος θα κατάφερνε ποτέ ακόμα και στην Ευρώπη να αντιποκριθεί σε τέτοια ανάγκη υποδομών. Ξέρουμε ότι η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ουσιαστικά δεν τα βγάζει πέρα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά οι τάσει αυτέ υπερβαίνουν τι δυνατότητέ τη και το αποτέλεσμα θα είναι ότι πολλά παιδιά θα μείνουν εκτός σχολείου, εκτός πανεπιστημίου, σε μια χώρα που πραγματικά έχει ανάγκη την παιδεία και την εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιες μπορεί να είναι δυσμενεί συνέπειε από την κατάσταση αυτή. Θέλουμε όμω να μπορούμε μέσω του προγράμματο αυτού να βοηθήσουμε κι εμεί και το θετικό νέο είναι ότι θα υπάρχει μια αύξηση πλέον του προσωπικού που θα μπορεί να δραστηριοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος αυτού. Δόθηκε και έγκριση από το Συμβούλιο. Θα μπορέσουμε λοιπόν εμείς να συνεισφέρουμε περισσότερο. Αλλά σε τι ακριβώς θα συνεισφέρουμε. Αυτό θα θέλουμε να το γνωρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ Σάρλε που μας το υπενθυμίσατε αυτό, γιατί ακόμα και αν έχουν την επιλογή απόκτησης παιδιών οι γυναίκες, τα παιδιά αυτά θα πρέπει στη συνέχεια να μπορούν να πάνε στο σχολείο και να μπορούν να απορροφηθούν από την κοινωνία. Η Ελένη θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βεβαίως, allow me to speak in Greek, my mother tongue. Μιλήσω στα ελληνικά, και μου γλώσσα. Uh, βεβαίως υπάρχει, έχω μια αιρετική ίσως άποψη για αυτό το ζήτημα με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι αυτός ο πλανήτης μπορεί να αντέξει ένα πληθυσμό πέραν των 7-6-7 δισεκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια και γι' αυτό γίνεται αυτή η αλυσιδωτή, τον domino effect από τη μια καταστροφή στην άλλη. Ακόμη και αυτές οι επιδημίες που εκδηλώνονται κατά καιρού είναι η αντίδραση της ίδιας της ε, φύσης στον υπερπληθυσμό και μη μου ζητήσετε τώρα να κάνω βιολογική προσέγγιση αυτού του ζητήματος. Είναι τεράστια σημασία να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό όσον αφορά το health and reproductive ε, education να ξέρουν με ποιο τρόπο θα αποκτήσουν ένα παιδί ή θα αποφύγουν μία εγκυμοσύνη είναι τεράστια σημασία ο οικογενειακό ε, προγραμματισμό. Είναι πολύ σωστό ότι με νόμου δεν μπορεί να ρυθμίσει αυτά τα ζητήματα. Δείτε στην Κίνα όπου είχαν επιβάλει το κότα του ενό παιδιού και γεννήθηκαν τώρα εκατομμύρια παιδιά τα οποία δεν έχουν καν ταυτότητα. Δεν υπάρχουν για τι αρχέ. Δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο όταν αρρωστήσουν γιατί δεν υπάρχουν απλώ. Δεν μπορούν να πάρουν ταυτότητα. Έχουν αποκρύψει από τι από ε, Το ίδιο συμβαίνει και σε ε, άλλα μέρη της Αφρικής. Έχουμε τα τρομερά εγκλήματα που γίνονται σε άλλες περιοχές, ειδικά με, την, με τις δολοφονίες νεογεννήτων μόλις, μόλις γεννηθούν τα παιδιά. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάση περισσότερο στον οικογενειακό προγραμματισμό και στην εκπαίδευση της κάθε γυναίκας και δεν μιλάμε για περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από δημογραφικές αλλοιώσεις. Για παράδειγμα, στη δική μου την πατρίδα ε, έχει πέσει δραματικά η, η γεννητικότητα στο κάτω από ένα παιδί ανά οικογένεια. Πολλοί δεν αποκτούν καν ε, παιδιά. Την ίδια στιγμή που γίνεται επικισμός από μια άλλη χώρα με τρομακτικούς ρυθμούς. Κάποια στιγμή δηλαδή θα βρεθούμε από την πλειοψηφία του 82% να είμαστε μια θλιβερή ε, μειοψηφία. Ε, μιλάμε για νορμάλ συνθήκες όπου δεν κινδυνεύει ένας λαός. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε τους ρυθμούς στο βαθμό που μπορεί να τους αντέξει μια κοινωνία ανάλογα με την ε, οικονομική της κατάσταση. Και η Κύπρος που είναι η πρώτη στην Ευρώπη ε, σε αυτό τον τομέα είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης. Κανείς δεν το γνωρίζει αλλά μάλλον να το βάλω πιο σωστά το gap μεταξύ των πάρα πολύ πλούσιων και των πολύ φτωχών είναι τεράστιο. Και οι πάρα πολύ πλούσιοι είναι ελάχιστοι και οι πολύ φτωχοί είναι η μεγίστη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Yeah, I think, um... Ευχαριστούμε. Κυρία Στένεκ, αναφέρθηκε σε αυτό το παράδοξο που υπάρχει σε κάποιες χώρες να υπάρχουν Πιέσει οικονομικέ προ τι γυναίκες, τις νέες γυναίκες να μην αποκτήσουν παιδιά. Και άλλε πιέσει εξαιτία του να μην μπορεί να βρει κανεί δουλειά, το, το, το κόστος της εκπαίδευσης του να βρει ε, σπίτι. Αυτό, αυτές τις πιέσεις τις διαπιστώνουμε κυρίως στη Νότια Ευρώπη, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως φαινόμενο εάν λάβει κανείς υπόψη του την ιστορία αυτών των χώρων. Κέβιν Μακάφη από ΤΕΦΚΟ, e μάλλον ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναπτυξιακή Συνεργασία. Νομίζω σας έχω ξαναδεί στην ομάδα μας. Ε, ε, θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι ακόμα στι ομιλήτριε. Αναφερθήκατε στη χρηματοδότηση από το UNFPA. Θέλω να σας ρωτήσω τι έγινε με τη χρηματοδότηση από τις Ηνωμένε Πολιτείες προς το πρόγραμμα του ΟΗΕ, το δικό σας. Τι συνέβη. Κύριος Μακάση. Ευχαριστώ και καλημέρα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση της έκθεσης. Είναι ενδιαφέρουσα. Χρειάζεται να γίνονται τέτοιες μελέτες για να ενημερωνόμαστε και να έχουμε επιχειρήματα. Πράγματι, ε, μία από τις προτεραιότητες μας είναι η βελτίωση των συστημάτων υγείας με ιδιαίτερη έμφαση στα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στη συνεργασία με τον ΠΟΗ για την ενίσχυση των συστημάτων υγεία που εστιάζεται ιδιαίτερα στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα. Θα ξεκινήσουν σύντομε σχετικέ προκηρύξει. Είναι μία από τι προτεραιότητε μα η εξασφάλιση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των κοριτσιών. Αυτό φαίνεται και στο κονσένσου για την ανάπτυξη και στο θεματολόγιο, καθώ επίση και την πρωτοβουλία του ΟΗΕ με το όνομα Spotlight. Πέρα από αυτό ε, έχουμε την υποστήριξη για συγκεκριμένες περιοχές, για την σχέση με την βία κατά των γυναικών και διάφορα εργαλεία. Και σε περιφερειακό επίπεδο υποστηρίζουμε λοιπόν και σε παγκόσμιο επίπεδο υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Το 2016 είχαμε μια χρηματοδότηση 470 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, αντίστοιχη σημαντική χρηματοδότηση πάνω το, άνω των 100 εκατομμυρίων ήταν στο πρόγραμμα Spotlight ε, και περίπου 100 εκατομμύρια για την υποσαχάρια Αφρική. Εδώ εστιάζουμε κυρίως στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες και τους νέους. Ένα άλλο ζήτημα είναι η πρόσβαση σε υπηρεσίες ε, οικογενειακού προγραμματισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εξετάσει το ζήτημα το, το, της α, πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες οικογενειακού ε, προγραμματισμού με χρηματοδότηση 20 έως 25 εκατομμύρια ε, για τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα το, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, στην τρέχουσα μάλλον προγραμματική περίοδο περιμένουμε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε περίπου 20-25 εκατομμύρια και βεβαίως γνωρίζετε ότι γίνεται η διαπραγμάτευση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα μεταβάσω το, τι ανησυχίε σας και τη συζήτηση που κάνουμε εδώ στου ανωτέρου μου για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τα μέσα που χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να καταφέρουμε να απευθυνθούμε ε, και να βοηθήσουμε όλες τις γυναίκες σε όλες τους τις ανάγκες. Αυτό δεν σημαίνει μόνο τα ζητήματα της υγείας, αλλά και ζητήματα όπως η εκπαίδευση, η πλήρης πρόσβαση στο, στις, στις υπηρεσίες υγείας και στον οικογενειακό προγραμματισμό αναδεικνύει η έκθεσή σας πόσο σημαντικό θέμα είναι η επιλογή. Αναφέρεται συχνά αυτή η λέξη. Βέβαια, το κρίσιμο είναι να δούμε πώς αυτό θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες δράσεις και να δούμε πώς τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συνεισφέρουν. Γνωρίζουμε ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα έχουν κρίσιμη σημασία για τη χειραφέτηση των γυναικών, θα έλεγα ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις αντίστοιχες του ΟΗΕ. Θα θέλαμε όμως επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και στο ζήτημα των σουξολικά μεταδεδομένων νοσημάτων ε, ε, και, και, και, επίσης την τη στηρότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταγράφουμε όλα αυτά τα οποία είπατε και ότι όντως τα ποσοστά γονιμότητα στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλά, όπως είπε και η Ελένη Θεοχάρους. Λοιπόν, ακούσετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω. Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας unfpa.org και βέβαια υπάρχουν και κάποια έντυπα αντίγραφα μέσα στην αίθουσα. Στο διαδίκτυο βέβαια είναι λίγο πιο διαδραστική εμπειρία, αλλά αξίζει να επισκεφτείτε την έκθεση και στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα όσα είπε ο κύριος Γκέρενς, η παγκόσμια πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία, τα σχετικά δικαιώματα, αποτελεί και μέρος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Τα όσα έθιξα λοιπόν σήμερα ήδη πριν από 50 χρόνια είχαν αναγνωριστεί ως αναπαραγωγικά δικαιώματα. Πάντως, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πλέον στηρίζουν πολύ στεναρά την προσέγγιση αυτή. Ουσιαστικά, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, ως προς τη συγκεκριμένη προθεσμία που έχει τεθεί, είναι μια προσπάθεια που προωθεί παράλληλα και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Και όπως είπατε και εσείς, ο οικογενειακός προγραμματισμός θα πρέπει να είναι καθολικά και παγκόσμια προσβάσιμος ως επιλογή και σε σχέση με τις παρατηρήσεις οι οποίες κάνατε και εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβαζα τις καμπύλες αυτές, τις γραφικές παραστάσεις τις οποίες σας παρουσίασα. Είναι εντυπωσιακή η μείωση, η πτώση στα ποσοστά γονιμότητος και γενετικότητος και αυτό έχει συμβεί πάρα πολύ γρήγορα σε ορισμένες χώρες και σε ορισμένες περιπτώσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση που έχει ριζώσει πια καλά Υπάρχουν σαφώ κάποιες χώρε με υψηλά ποσοστά γενετικότητας, αλλά αποτελούν πλέον την μειοψηφία. Υπάρχουν κάποιες χώρε στην υποσαχάρη Αφρική, ο Νίγηρας για παράδειγμα, αλλά και χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή χώρες οι οποίες ταλανίζονται από συγκρούσεις ή γενικά άλλους παράγοντες που βάλουν κατά των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Ευπαθείς ουσιαστικά χώρες που δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των ανθρώπων και που δεν καταφέρνουν τελικά να δώσουν απαραίτητη πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, φροντίδας κτλ. Όσον αφορά το δικό σας ερώτημα, Πρόεδρε, για τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού από τα Ηνωμένα Έθνη, από τις Ηνωμένε Πολιτείε, μάλλον. 70 εκατομμύρια ετησίως ήταν η πρικοδότηση από τις Ηνωμένε Πολιτείε στην περίοδο Ομπάμα. Με τη νέα όμως τώρα κυβέρνηση στις Ηνωμένε Πολιτείε, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί. Πρέπει να σας πω επίσης ότι αυτό συνέβαινε όμως και με άλλες κυβερνήσει ρεπουμπλικανών στι Πολιτείε. Γενικότερα η χρηματοδότηση ήταν πιο υψηλή όταν είχαμε δημοκράτε μάλλον προέδρους από τους δημοκρατικούς. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ θετικό αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά την ακούσια, την ανεπιθύμητη γονιμότητα, εγκυμοσύνη. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί και θέμα δημόσιας πολιτικής για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέπουν την ακούσια εγκυμοσύνη την επιθύμητη γονιμότητα, η οποία μπορεί ουσιαστικά να συνδέεται ακόμα και με τα STIs, δηλαδή τις ε, σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και αυτές οι πολιτικές πρόληψεις και έπειτα πρέπει να υπάρχουν και πολιτικές για τα ζευγάρια εκείνα τα οποία δεν μπορούν για τον έναν τον άλλο τρόπο να συλλάβουν. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα προγράμματα για να βοηθούν τα ζευγάρια αυτά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα παιδί, να προβλέπεται χρηματοδότηση και για αυτού του είδου τι δημόσιε πολιτικέ, οι οποίες σε κάθε περίπτωση μπορούν να έχουν μια πολύ σημαντική συμβολή. Τώρα, η παγκόσμια καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και αναφερόμαστε εδώ πέρα και στα μέτρα αντισύλληψης, θα πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο ενισχύει τα ατομικά δικαιώματα, το οποίο να μην επιτρέψει σε καμία περίπτωση διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών ή του αναγκαστικού γάμου, καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση για τα γόρια και τα κορίτσια, τα οποία να μπορούν κατά αυτόν τον τρόπο να προετοιμάζονται πολύ καλύτερα όσον αφορά τι αποφάσει που θα χρειαστεί αργότερα να πάρουν στη ζωή του. Και βέβαια στι αποφάσει αυτέ θα πρέπει να περιλαμβάνονται και όλε αυτέ οι αποφάσει που έχουν να κάνουν με την αναπαραγωγική υγεία. Και έχουμε και κάποιε χώρε όπου το κοινωνικό πρότυπο προβλέπει πολύτεκνες οικογένειες, πολυπληθείς οικογένειες. Και βέβαια στις περιπτώσεις αυτές έχουμε γυναίκες οι οποίες έχουν αποκτήσει περισσότερα παιδιά από ό,τι θα επιθυμούσαν πραγματικά. Είναι σημαντικό στις χώρες αυτές, για παράδειγμα στη Ρουάντα, να υπάρχουν οι απαραίτητε καμπάνιε, οι απαραίτητε εκστρατείε. Στη Ρουάντα είχε γίνει αυτό τα τελευταία χρόνια και τώρα και οι ίδιοι άντρε προτιμούν μικρότερη οικογένεια, λιγότερα παιδιά από ό,τι γυναίκε πολλέ φορέ. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ όλος ιδιαιτέρως ε, την υποστήριξη που δεχόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό. Όντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ όσον αφορά το ζήτημα της προϊκής υγείας και των σχετικών δικαιωμάτων και η υποστήριξη που λαμβάνουμε για το Ταμείο μας πραγματικά επιτρέπει τελικά σε πάρα πολλές γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη εφόσον το επιλέξουν. Και η πρωτοβουλία Spotlight επίση είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο από χρηματοοικονομικής πλευρά, ακριβώ επειδή υπάρχει όλη αυτή η σημαντική πρικοδότηση, αλλά κυρίω ακριβώ επειδή ευαισθητοποιεί πάρα πολύ του πολίτε για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών και συμβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν όλε αυτέ οι δυσμενεί πρακτικέ κατά των γυναικών. πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πολύ για την έκθεση αυτή και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά ότι όντω υπάρχει απαραίτητη υποστήριξη και τα προγράμματα αυτά που δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέγουν πραγματικά όσον αφορά την τα ζητήματα αγωνιμότητος. Ας περάσουμε τώρα στα σημεία 22 και 23 της ημερήσια διάταξης, εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με το ΦΛΕΚΤ, την επιβολή της δασική νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο. Ο Γιάννα Ζαραντήλ θα κάνει κανονικά την παρουσίαση, η Ελένη και ο Κάρλος όμω θα μα κάνουν την παρουσίαση, η Ελένη Θεοχάρου, με συγχωρείτε θα μα κάνει την παρουσίαση. Ξέρετε ότι πέρυσι είχαμε στείλει στο Καμερούν μια αποστολή προκειμένου να παρακολουθήσουμε εκεί το πώς εφαρμόζεται το FLECT. Και τον Ιούλιο εγκρίναμε μια έκθεση για την λογοδοσία και την υπεύθυνη διαχείριση των δασών και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια εγκρίναμε το ψήφισμα αυτό. Τώρα επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο Βιετνάμ. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν προχωρήσει σε μια εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση προκειμένου όλες οι εισαγωγές ξυλίας από το Βιετνάμ να είναι ουσιαστικά εισαγωγέ προϊόντων που έχουν αποκτηθεί με τον πλέον νόμιμο τρόπο. Και ξέρετε ότι αντίστοιχε πρωτοβουλίε είχαμε και σε άλλου τομεί, όπω για παράδειγμα τα ορυκτά και η εξόριξη ορυκτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να παρακολουθούμε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Θα δημιουργηθεί λοιπόν πλέον ένα σύστημα το οποίο θα εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία για το ΦΛΕΚΤΑ, δηλαδή που θα προβλέπει την επιβολή τη Ευρωπαϊκή Δασική Νομοθεσία για τα προϊόντα αυτά τα οποία θα φτάνουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι σημαντικό λοιπόν να επικυρωθεί η εθελοντική αυτή συμφωνία εταιρική σχέση. και Εμεί καλούμεθα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μα και θα υποβάλουμε και μία πρόταση ψηφίσματο και για την πρόταση ψηφίσματος αλλά και για τη σύμφωνη γνώμη εμείς γνωμοδοτούμε ως Επιτροπή ανάπτυξη. Η Ελένη Θεοχάρους λοιπόν έχει και πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Chair Lady. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, ο συνάδελφος ο Γιάννης Χραντήλ δεν μπορεί να είναι μαζί μας εδώ σήμερα, αλλά θα παρουσιάσω εγώ την έκθεσή του Πρώτα να τονίσω ότι ο Γιάννης ο εισηγητής μας στην Διεθνή Επιτροπή Υπάρχει σύνδεση με την Επιτροπή αυτή επί της ουσίας και μπορεί να φέρει περισσότερη συνογή, συνέργειες και εμπειρογνωμοσύνη στην μελέτη αυτή του εγγράφου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινή ευθύνη για την υποβάθμιση των δασών όχι μόνο επειδή προϊόντα που σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες εισάγονται στην αγορά μας η ξυλία είναι το μόνο προφανές αλλά όχι το μόνο παράδειγμα υπάρχουν και άλλα προϊόντα όπως ε, το φινικέλαιο τα οποία και αυτά εμπλέκονται στη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, και την πρωτοβουλία για το FLECT. Εξάγει σε χώρες ε, στις οποίες εμπλέκονται διάφοροι, διάφορα ενδιαφερομένα μέρη όπου θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, σωστά η νομοθεσία. Ο έλεγχος της προμήθειας και της νομιμότητας του συστήματος ε, περιλαμβάνει πιστοποίηση της νόμιμης ξυλίας πριν την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Η εταιρική σχέση μεταξύ της Ένωσης και της αντίστοιχης χώρας μας δείχνει το πώς θα πρέπει να λειτουργεί όλο αυτό. Η επιτυχία τη της πρωτοβουλία ΦΛΕΚ θα εξαρτηθεί από την ε, αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βιετνάμ είναι ε, από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ε, ξύλες και άλλων δασικών προϊόντων στον κόσμο. Είναι ηγέτης, ε, είναι πρώτη επίσης στην εξαγωγή επίπλων. Έχει συμμεθεί μεγάλη βελτίωση στην διαχείριση των δασών. Έχει διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συμφωνία FLEGT η έγκριση και η θέση σε ισχύ αυτής της συμφωνία ε, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου. Ο συνάδελφος μου Γιάννη υποστηρίζει ε, την διαδικασία φλέκτ με το, ε, με το Βιετνάμ. Θα ήθελε το ψήφισμα να δώσει έμφαση σε τρία σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε. να σταματήσει παρά, η εισαγωγή παρά ξυλία από γειτονικέ χώρες Πολλές από τις 3.000 εταιρείε που εργάζονται στην ξυλία ε, στο Βιετνάμ εξαρτώνται από την εισαγωγή ξυλίας από το Λάος και την ε, Καμπότζη. Ε, η εκμετάλλευση των πόρων τα τελευταία χρόνια είναι υπό όπως θα έπρεπε να είναι και σε κάθε άλλη περιοχή στο Λάος είναι παρκής στην παρακολούθηση, στην Καμπότζη χρειάζεται να βελτιωθεί. Το δεύτερο σημείο του Βιετνάμ έχει δεσμευτεί να συμπεριλάβει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ε, εφαρμογή της συμφωνίας υπάρχει μια ομάδα που έχει ε, ιδρυθεί από την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει 29 οργανώσεις από τις ενώσεις εργαζομένων στον τομέα της ξυλίας, ε, επιχειρηματιών, ε, δικαιούχων του ΦΛΕΚΤ και διάφορα, διάφορους άλλους οργανισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χνηλασιμότητα ως προς την προέλευση ε, της ξυλίας. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ θα πρέπει να αναπτύξει περισσότερες μεθόδους συνεργασίας ώστε να υπάρξει διαφάνεια και γρήγορη ε, διαβίβαση των εγγράφων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να υπάρξει υποστήριξη στο πρόγραμμα και να υπάρξει επίσης παρότριση ε, προς τα κράτη-μέλη την εφαρμογή του προγράμματος. Θα στείλουμε ε, το μήνυμά μας και στην ε, Επιτροπή, Επιτροπή, την ε, Ίντερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν γνωρίζω αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι συμφωνώ με αυτή τη συμφωνία που θα είναι μια σημαντική συμβολή στην ε, εξάλληψη της παράνομης εισαγωγής ε, ξυλίας. Όσον αφορά προηγούμενες συμφωνίες με χώρες στην Αφρική και στην Ινδονησία, βασίζονται στην ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό τη σημαντική συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών ε, και θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή τη νομοθεσίας ε, τη συμφωνίας αυτής. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι οι ε, ντόπιε κοινότητε βασίζονται πάρα πολύ στην, στον κλάδο της ξυλίας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις δεσμεύσεις μας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν θα πρέπει να δούμε αυτή τη συμφωνία ως ε, ε, ένα μέσο για να εκμεταλλευτούμε τους δασικούς πόρους. Θα πρέπει να ε, αποτρέψουμε την... Αποδάσει που λαμβάνει χώρα και στην Ευρώπη και επίσης να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε επιτυχώς να παρακολουθήσουμε τον αντίκτυπο της ε, συμφωνίας. Θα πρέπει φυσικά η Επιτροπή να δίνει αναφορά στο Κοινοβούλιο για την εφαρμογή. <clears throat> Κύριε Γκέρενς, εγώ έχω μια ερώτηση τεχνικού χαρακτήρα προς την Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία για την πιστοποίηση των δασών προβλέπει δύο. Πιστοποιητικά FSA και ε, FTA είναι λίγο τεχνικό και τα δύο επιδιώκουν την βιώσιμη ανάπτυξη των δασών και γνωρίζω ότι έχουμε αυστηρούς κανονισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ξυλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ε, απλά λόγια πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το σύστημα. Γνωρίζω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να τηρήσουν όλους τους κανόνες για να εισαγάγουν ξυλία, όμως είναι περίπλοκη η νομοθεσία και κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε για τη συμφορία για μια άλλη χώρα σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να δεχόμαστε ξυλία από, μια, από ένα δάσο το οποίο δεν έχει πιστοποίησης Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ψήφισμα μας δίνει την δυνατότητα να εξηγήσουμε ποιοι θα είναι οι όροι που θα πρέπει να τηρηθούν από το Βιετνάμ. Θα ήθελα να σας θυμίσω κάποια σημαντικά σημεία από την πλευρά των πρασίνων θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική ε, τήρηση των υποχρεώσεων, να υπάρχει ιδέουσα επιμέλεια και να υπάρχουν δεσμευτικοί όροι στην αλυσίδα ε, εφοδιασμού. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής παράνομης ξυλίας στην αγορά του Βιετνάν. Να υπάρξουν δηλαδή δεσμευτικές διατάξεις και να υπάρξει και ένας μηχανισμός κυρώσεων παράλληλα. Thing, uh, Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσει το Βιετνάμ για το επόμενο α, προγραμματισμό να δεσμευτεί, κάνετε λόγο για την συμμετοχή της κοινωνίας των ε, πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό σημείο και αυτό το να μπορούμε να λαμβάνουμε πληροφορίες και από ανεξάρτητες πηγές. Και τέλος θα πρέπει το Βιετνάμ να αντιμετωπίσει το θέμα της διαφθοράς. Αναφέρουμε στο σκάνδαλο του Rosewood, του συγκεκριμένου τύπου ξυλίας, να σταματήσει παράνομη εισαγωγή ξυλίας από την ε, Καμπότζη Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπω θέλει να απαντήσει σε ερωτήσει που ακούσαμε. Δεν έχω το όνομά σα δυστυχώ, Πείτε μα ποιο είστε. δυστυχώ δεν έχω το όνομά σα, λέει ο Πρόεδρος. Λουκα Περέθα. Από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Όντως, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξέφρασαν τις απόψεις τους για το ζήτημα αυτό. Καταρχάς, είμαστε υπέρ της ισχυρής υποστήριξης που εκφράσατε για τη συμφωνία αυτή, τόσο ο εισηγητής όσο και οι προαγλήσαντες. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο παρελθόν, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ θα αποβεί τελικά μια πολύ σημαντική συμφωνία η οποία θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Τονίστηκε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική συμφωνία αυτή για την παγκόσμια αγορά, για τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού, γιατί αναφερόμαστε εδώ πέρα σε 80 τρίτες χώρες, εκ των οποίων ορισμένες κινδυνεύουν ε, από παράνομη υλοτομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή και η αξιόπιστη στεναρή εφαρμογή της όντως θα αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Από αυτή την οπτική λοιπόν γωνία θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία έθιξαν οι ευρωβουλευτές. Πρώτον, να σε υπενθυμίσω ότι το BPA, η συμφωνία αυτή προβλέπει ένα πλήρε νομικό πλαίσιο για την εμπορία ξυλίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Υπενθυμίζει όμως ότι η συμφωνία καθώς επίσης και το σύστημα εγγύησεων θα καλύπτει όλες τις εξαγωγές από το Βιετνάμ. Δεν θα ασχοληθούμε λοιπόν μόνο με τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική αλυσίδα εφοδιασμού, αλλά με όλο τον κλάδο και τις εξαγωγές που ο κλάδος αυτός προωθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η πρόοδο όσον αφορά την βιώσιμη διαχείριση των δασών του Βιετνάμ είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί και τονίζεται συμφωνία. Η προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα πλήρη και συνδέεται και με άλλε προσπάθειε που έχουν γίνει για την διατήρηση των δασών στη χώρα, όπως και η εφαρμογή των όσων προβλέπονται για τα δάση στα πλαίσια της Σύμβασης για το κλίμα. Και επίσης αναφερόμαστε εδώ πέρα και στις συγκεκριμένες εισαγωγές Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό μα απασχόλησε πάρα πολύ στι διαπραγματεύσει που είχαμε με το Βιετνάμ και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τώρα η κυβέρνηση του Βιετνάμ στα πλαίσια του BPA μα λέει ότι θα υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανή, μηχανισμοί εφαρμογή οι οποίοι θα βασίζονται σε ένα μηχανισμό μελλοντική νομοθεσία όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, που θα ευθυγραμμίσει τελικά το νομικό πλαίσιο του Βιετνάμ με αυτό το οποίο ήδη υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια ακόμα πρέπει να καταβάλουμε πολλές προσπάθειες προκειμένου να εφαρμόσουμε όλες τις διαφορετικές πτυχές αυτής της συμφωνίας, όπως ξέρουμε και από άλλες τέτοιες συμφωνίες, θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για να γίνει αυτό, διότι θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του σχετικού πολιτικού πλαισίου, θα πρέπει να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν απαραίτητε ικανότητες σε διάφορα επίπεδα και θα πρέπει από κοινού με το Βιετνάμ να καταφέρουμε να επαληθεύσουμε ανεξάρτητα την ετοιμότητα για να ξεκινήσουν οι άδειε FLECT και να δούμε τελικά αν μπορούμε όντω να εφαρμόσουμε τα κριτήρια τα οποία διέπουν τη συμφωνία αυτή. Να αναφερθώ και σε κάποια άλλα σημαντικά ζητήματα που έθιξαν ο εισηγητέ αλλά και άλλοι βουλευτές, το ζήτημα των, της εμπλοκής των ενδιαφερομένων μερών. Και αυτό είναι μια σημαντική πτυχή τη εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέση, αλλά και γενικότερα τη πρωτοβουλία ΦΛΕΚΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδο και βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεσμεύεται πλέον με τον, με την κοινότητα των πολιτών και με τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή αυτή τη συμφωνία. Θεωρούμε ότι η διαδικασία συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι μια διαδικασία η οποία εξακολουθεί και ισχύει και υπάρχει μια γενικότερη δέσμευση προκειμένου να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης, αλλά και στην εφαρμογή της ίδιας συμφωνίας. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι έχει ήδη γίνει σημαντική εργασία όσον αφορά την προετοιμασία της εφαρμογής συμφωνίας. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ έχει ήδη εφαρμόσει διάφορες νομικέ μεταρρυθμίσει, μια νέα δασική νομοθεσία για παράδειγμα, που ήδη προβλέπει ορισμένες από τι κέρυε διατάξει συμφωνίας αυτή προκειμένου όντω να καταφέρει η κυβέρνηση του Βιετνάμ να εφαρμόσει πλήρω την Εθελοντική Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Η συμφωνία αυτή αποτελεί όμω μόνο μέρο τη πολιτική μα για την καταπολέμηση τη παράνομη υλοτομία. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοτομία και όπως θα έχετε δει και από την έκθεση για την διετή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής που πρόσφατα δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί πέρα όπως βλέπετε επικεντρωνόμαστε στην ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί από τότε που το Μάρτιο του 2013 σε ισχύ η νέα αυτή νομοθεσία αλλά βρίσκονται όλα ακόμα σε εξέλιξη, καθότι θέλουμε να εφαρμόσουμε πλήρως και αυτή τη νέα αρχή της δέουσας επιμέλειας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετέθη επίσης ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τον ρόλο των, συστημάτων ε, ιδιωτικής αδειοδότηση Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να απαντηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού για την υλοτομία του νομικού αυτού πλαισίου. Προβλέπεται λοιπόν αυτό το ιδιωτικό σύστημα διοδότηση για του φορεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι πλήρω ενήμεροι για όλου του κινδύνου που μπορεί να υπάρχουν ω προ την νομιμότητα τη διαδικασία υλοτομία. Τώρα, η αδειοδότηση δεν είναι ε, υποχρεωτική απέτηση στα πλαίσια της κοινοτικής αυτής νομοθεσίας για την ξυλία. Παρόλα αυτά, η παροχή άδεια μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους διάφορους φορείς οικονομικής εκμετάλλευση. Δηλαδή, προβλέπεται ότι μέσω του συστήματος αυτού θα γίνονται απαραίτητε επαληθεύσει κινδύνου, η απαραίτητη αξιολόγηση κινδύνου. Καλείται δηλαδή ο φορέα να δει αν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος στην όλη αλυσίδα εφοδιασμού όσον αφορά την υλοτομία, να είναι δηλαδή παράνομη. Και θα πρέπει επίσης να καλύπτεται μέσω της αδειοδότησης αυτής όλες οι πτυχές νομιμότητας που προβλέπει η νομοθεσία και να μην προκύπτει καμία ανησυχία για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας επί τόπου. Γιατί ξέρετε πολύ συχνά είναι πολύ μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στο τι προβλέπεται από ένα πρότυπο σε μια κοινοτική νομοθεσία και τι γίνεται στην πράξη επί επιτόπου σε συγκεκριμένες χώρες ή σε συγκεκριμένε περιστάσει. Έχω καταγράψει τι υπόλοιπε παρατηρήσει που γίνανε από του προλαλήσαντε και θεωρώ ότι όλα αυτά θα ενταχθούν ούτως ή άλλως στη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας και θα διαμορφώσουν τελικά και την πρόταση ψηφίσματος την οποία θα εγκρίνει η Επιτροπή Ίντα. Και βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεσή σα προκειμένου σε τακτική βάση να σα δίνει πληροφορίε για τη μελλοντική εφαρμογή τη συμφωνία αυτή και βέβαια θα είμαστε στη διάθεσή σας ε, για να ε, μεταφέρουμε προς την κυβέρνηση του Βιετνάμ και τα όσα είπατε στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ελένη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι 11 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία 21 και 22 Ιανουαρίου. Το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε έχει σχέση με τη ζάχαρη. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να συζητήσουμε να κάνουμε ένα ε, μικρό πεντάλεπτο διάλειμμα για να ετοιμαστούν οι επόμενοι μιλητές. Okay, colleagues, we can resume now item which is item... Αγαπητοί συναδελφοί, ας περάσουμε στο σημείο 24 της μερίσιας διάταξης, προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδοτήσεις για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, συνέπειες για τους παραγωγούς ζάχαρης στις χώρες ΑΚΕ. Προβλέπεται εδώ πέρα μια ανταλλαγή απόψεων με τον Τίλα Βέρνον, πρέσβη τη Μπελίζε, ο οποίο παράλληλα και πρόεδρο τη Υποεπιτροπή των Χωρών ΑΚΕ για τη Ζάχαρη. Ξέρω ότι το ζήτημα αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλοί ευρωβουλευτέ στο παρελθόν έχουν προσπαθήσει να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στου παραγωγού ζάχαρη στι χώρε εταίρου. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο προβλέπεται η σημερινή ανταλλαγή απόψεων είναι για να μιλήσουμε περισσότερο για τα ζαχαρότεπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ο εφιστάμενο καονισμός τη κοινή γεωργική πολιτικής προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο συνδυασμένη υποστήριξη για συγκεκριμένε μορφέ καλλιέργεια στις οποίες περιλαμβάνεται και ο τομέας των ζαχαρότευτων. Στόχος λοιπόν του μέτρου αυτού είναι τα κράτη-μέλη να έχουν το απαραίτητο περιθώριο ευελιξία και να καταφέρουν να συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των αγροτικών εισοδημάτων. Αυτό μάλιστα απαιτείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω δει, 11 κράτη-μέλη έχουν παράσχει μια θελούσια συνδυασμένη υποστήριξη στον τομέα των ζαχαρότευτών. Θυμάμαι ότι στο παρελθόν, στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής, προσπαθούσαμε να δούμε αν θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην επόμενη γεωρική πολιτική μηχανισμή αυτή. Τώρα, από, σε μια επιστολή της 11ης Οκτωβρίου 2018, ο πρέσβης Βέρνον Μα εξήγησε ότι οι χώρε ΑΚΕ θεωρούν ότι η εθελούσια αυτή συνδυασμένη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα επιζήμια όσον αφορά την παραγωγή ζαχαρότευτλων των κρατών ΑΚΕ. Είναι λοιπόν μαζί μας ο πρέσβης Ντίλαν Βέρνον για να μας μιλήσει περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ΑΚΕ αντιλαμβάνονται το σύστημα αυτό εθελούσα συνδυασμένης υποστήριξης από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Κύριε πρέσβη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα Μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδελφοι από τα κράτη-μέλη, τα κράτη της ΑΚΕ. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή ε, της ΑΚΕ για την ζάχαρη αντέδρασε άμεσα στην επιστολή όπου εκφράσαμε την ανησυχία μας για την προοδευτική συνδεδεμένη στήριξη συγκεκριμένα στον τομέα της ζάχαρης και που οδήγησε στην πρόσκλησή μα εδώ. Η ζάχαρη συνεχίζει να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο κοινωνικό και οικονομικό στις χώρες της ΑΚΕ και κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμένες και είναι πολύ σημαντική ως προς την επίτευξη των ε, βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων. Ε, έχει μια επίπτωση ε, πολλαπλασιαστική στις οικονομίες όπου και οι εταιρείε έχουν πολλά ωφέλη. Η έκθεση που εκδόθηκε το 2016 που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ομάδα για τις χώρες ΣΑΚΕ αναφέρει ότι είναι βασικός μηχανισμός η βιομηχανία της ζάχαρης ε, για ε, τις χώρες της ΑΚΕ. Από το 2006 κατέστησε σαφές η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι το καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση ώστε ε, οι αγρότες να ανταποκρίνονται στις ε, τιμές της αγοράς. Η τιμή αναφοράς για τη ζάχαρη λοιπόν μειώθηκε ε, από 632 ευρώ ανατόνο σε 400 ευρώ ανατόνα και καταργήθηκε η ελάχιστη τιμή τον Οκτώβριο του 2017 όπως γνωρίζουμε. Η, η, τιμή που ορίστηκε για το 2018 ήταν 3, 347 ευρώ ανατόνο. Πολλές χώρες βέβαια έχουν πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο αναμένοντας αυτή την ανταγωνιστική εμπλοκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2006 αφιέρωσε 5,2 εκατομμύρια ευρώ για τον κλάδο της ζάχαρης και οι χώρες της ΑΚΕ που συμμετείχαν στο πρωτόκολλο έλαβαν 1,2 εκατομμύρια. Τα πρωτόκολλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί μπορούν και με τους ε, εχώριους πόρους οι βιομηχανίες της ζάχαρης έχουν την ευκαιρία να ε, επιβιώσουν σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Όμως, απρόσμενα, χωρίς διαβουλεύσεις, όπως ε, προβλέπεται από τα άρθρο 12 της Συμφωνίας του Κοτονού, και ενάντια στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015 και το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση εφάρμοσε προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για τα τσαχαρατεύτλα. Είναι μια επιδότηση για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση των χωρών ΑΚΕ, μιλάμε για 300.000 εκτάρια σε 11 κράτη-μέλη. Έχοντας υπόψη την ανάγκη που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 18 εκατομμύρια τόνους, θεωρούμε ότι, είναι πολύ ε, ε, θεωρούμε ότι υπάρχει διαστρέβλωση της αγοράς με αυτή την προαιρετική συνδεμένη στήριξη. Οι απώλειες εξαιτίας της συμφωνίας ανέρχονται στα 20 εκατομμύρια ετησίω. Αυτό είναι το ελάχιστο. Διατηρώντας την παραγωγή της ζάχαρης που δεν θα υπήρχε οι συμφωνίε αυτές κατά την άποψή μα. παρόλο που μπορεί να επενούνται μειώνουν το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές μειώνει τις τιμές, απειλεί τις εναλλακτικές αγορές ε, για τις χώρες της ΑΚΕ και είναι σε αντίθεση φυσικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη συνοχή και την ανάπτυξη. Επίσης αυτό είναι αντίθετο στις διαβεβαιώσεις που έχουν ε, δοθεί στις χώρες ΑΚΕ ότι ένα επίπεδο προτίμηση θα διατηρηθεί για την, προ... για την από τις χώρες της ΑΚΕ εξαιτίας των επενδύσεων που έχουν γίνει ώστε να υπάρξουν οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις στις ε, αντίστοιχες ε, βιομηχανίες. Γι' αυτό σας καλούμε κυρία Πρόεδρε να σταματήσετε και να καταργήσετε ε, τις προεδρικές συνδεμένες στήριξη στον τομέα της ζάχαρης και να βρείτε έναν τρόπο να αντιμετωπίσετε την τρέχουσα κατάσταση. Έχουν συμβάλει φυσικά την αύξηση των εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σύμφωνα με την εξελίξη που σας παρουσιάζουμε εδώ κάποιοι παραγωγοί δεν θα ήταν παραλόγο να ζητήσουν και αποζημίωση. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε εμπλεξεί και τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη δικιά μας οπτική δεν υπάρχει πρόθεση να εξεταστούν εντελεχώς ε, οι επιπτώσεις των συμφωνιών αυτό στην αγορά της ζάχαρης ο Επίτροπος, ο Αρμόδιος, σε σχέση με την ε, συνοχή της πολιτικής, έκανε αναφορά στην προστασία των προτιμήσεων. Ε, ως μέλος της ε, κοινής ε, κοινοβουλευτική συνέλευση ε, μεταξύ Χρόνα και, και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω ανυπόμονα ε, την ε, ανταπόκρισή σας. Η Υποπιτροπή για τη Ζάχαρη είναι πολύ ε, κοντά στην Επιτροπή σας όσον αφορά τις ε, στις χώρες της ΑΚΕ. Αναμένουμε την παρέμβασή σας να μας βοηθήσετε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να διασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία της Σάχαρης στις χώρες της ΑΚΕ θα παραμείνει βιώσιμη και ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες αυτές και με την κατάργηση των προαιρετικών συμφωνιών στήριξης θα μπορέσει να υπάρξει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Um, thank you, thank Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσει και η Γενική Διεθνήση Άγκρη. Για Σαλγκόνς. Σας ευχαριστώ. Περισσότερο παρατήρηση είναι παρά ερώτηση. Εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει την πορεία των διαπραγματεύσεων θα θυμούνται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Βραζιλίας είχε υπεραμεινθεί του, του δικαιώματος της προστασίας και θα έλεγα ότι αυτό ήταν που είχε δημιουργήσει μια κάποια ενόχληση και δυσκολία στι σχέσει μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή προφανώ είχε ε, ε, θετικά στοιχεία για τι χώρε ΑΚΕ και εγγυάται ένα επίπεδο τιμών και αυτό οδήγησε στην παρέμβαση ορισμένων χωρών, όπως για παράδειγμα η Βραζιλία, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ζάχαρης. Θα έλεγα ότι είναι αυτές οι αναδυόμενες οικονομίες που τα κατάφεραν να μας διχάσουν. Ε, θεωρώ εγώ ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των χωρών ΑΚΕ ήταν γενναιόδοροι. Και δεν θα έλεγα ότι είναι οι χώρε ΑΚΕ εκείνε οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν. Ε, αντιθέτως. Ε, βέβαια δεν πρέπει κανεί να είναι έτσι α, ε, Βλέπουμε μια συστηματική επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποτεδήποτε χρησιμοποιεί γενικευμένες προτιμήσεις για να αλλάξουν ουσιαστικά την κατεύθυνσή μας όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο. Πιστεύω ότι ε, η Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Συνεργασία πρέπει να πούμε ότι πρέπει να προστατεύεται ο πιο αδύναμος και να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιεί τους μηχανισμούς που έχει για προς αυτό. Βλέπουμε λοιπόν μια τάση την οποία κανείς πλέον δεν καταφέρνει να ανακόψει και πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αφενός τα πλεονεκτήματα που οι γενικές, γενικές προτιμήσεις μας έχουν δώσει, αφενός, και αφετέρου να βρούμε εναλλακτικέ ε, έτσι ώστε να αποζημιωθούν εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις εξέλιξεις. Ε, εναλλακτικέ, για παράδειγμα, για ε, τις χώρες ΑΚΕ, για χώρες στην Αφρική που έχουν επιχειρήσεις επεξεργασίας ζάχαρης. Είναι δύσκολη αυτή η διαπίστωση, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν θα χρειαζόταν να γίνει ή δεν θα είχαμε οδηγηθεί στο αδιέξοδο εάν γινόταν η συζήτηση άλλη εποχή. Μαξέλεση. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσει κανείς για την αθεώρηση της ΚΑΠ και σε σχέση με την σχέση μας με άλλες τρίτες χώρες. Για τους πράσινους, ο στόχος θα πρέπει να είναι διατροφική ασφάλεια, έτσι ώστε και, αυτό να το επιτύχουμε μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν στις μικρές εκμεταλλεύσεις αυτές οι επιλογέ. Θα πρέπει να λάβουμε υπέψουμε στο δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στην ανάπτυξη, το οποίο σημαίνει ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να μην οδηγεί στο ντάμπικ, να μην οδηγεί στην αρπαγή γεών και τέτοιου τύπου προβλήματα. Ξεκινώ έτσι για να δούμε το πρόβλημα στο σύνολό του. Μετά πρέπει να σκεφτούμε διάφορες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Πράγματι, η ζάχαρη είναι ένας ευαίσθητος τομέας, αλλά δεν είναι ο μόνος. Έχουμε και το, το βαμβάκι ή τα γαλακτοκομικά. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει μια εξάντεξιολόγηση των στηρίξεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι στηρίξεις δεν προκαλούν βλάβη, ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα δικαιολογημένη κοινωνική ανάγκη, την οποία να μπορούμε να αποδείξουμε με στοιχεία και Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι αυτή η στήριξη δεν δημιουργεί ε, στον ανταγωνισμό ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό και ότι πραγματικά βοηθάει τη διατροφική μας ασφάλεια. Έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, δυσμενείς συνέπειες για την αγροτική βιομηχανία στις τρίτες χώρες. Επίσης, πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να δίνεται στήριξη σε αγορές όπου η κρίση έχει προέλθει από υπερπαραγωγή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημα είναι αν οι συνδεδεμένες στηρίξεις θα πρέπει να μειωθούν ή και να καταργηθούν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις αναπτυσσόμενες χώρες, εκείνες, όπου διαπιστώνεται ότι οι συνδεδεμένες στηρίξεις δημιουργούν προβλήματα στην αγορά τους για να ληφθούν ε, μέτρα τα οποία θα αντισταθμίζουν τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητάει άλλο συνάδελφο το λόγο. Κύριο Νιά, εάν το προφέρω σωστά, η κυρία, συγγνώμη. Μάικλ, εντάξει. <laughs> δεν, δεν είμαι αυτό το πρόσωπο, λέει ο μιλητής. Πείτε μας ποιος είστε το λέει η πρόεδρος. Βαγγέλη Νεκράσιου από την Γενική Διεύθυνση Γεωργία από το διεθνε τμημα Τμήμα, Μονάδα 1α. Ασχολούμαστε εκεί πέρα με τι χώρε ΑΚΕ και ιδιαίτερα εγώ με το ζήτημα τη ζάχαρη, τη δική μου τη μονάδα. Προκειμένου να σχολιάσω τα όσα υπόθηκαν αυτή τη στιγμή για τη ζάχαρη και τι χώρε ΑΚΕ. Καταρχάς, ποια είναι η απόψή μα και η δική μα η αξιολόγηση όσον αφορά το συγκεκριμένο αυτό μέτρο για την προαιρετική στεδεμένη στήριξη και το πώς επηρεάζει τελικά τις χώρες ΑΚΕ σε σχέση με την παραγωγή ζάχαρης. Εμείς θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο αυτό μέτρο έχει ένα πολύ περιορισμένο προπολογισμό και πεδίο εφαρμογή. Μόνο στόχος του μέτρου αυτού είναι να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγής, κυρίως στους πιο ευαίσθητους τομείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής πλευράς και από κοινωνικής πλευράς. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μόνο σε 11 κράτη-μέλη και τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία έχουμε δεν δείχνουν ότι υπάρχει κάποια αντιστοίχηση με την εφαρμογή του μέτρου αυτού και το συνολικό ποσό ζάχαρης ή συγκεκριμένα καλλιέργειας ζαχαρότευτλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η επιπτώση από την εφαρμογή της προληπτικής δεδεμένης στήριξης είναι πολύ περιορισμένη και δεν οδηγεί σε στρέβλωση. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο νίκει στο μπλε κοιτίο, το blue box του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνάδει με τους κανόνες του ΠΟΕ δηλαδή, και θεωρούμε ότι χάρη στο μέσο αυτό, μάλλον εξαιτία του μέσου αυτού δεν επηρεάζεται ο γενικότερος σχέλισμό παραγωγή ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν οδηγεί σε μείωση για τις χώρες εκείνες που εφαρμόζουν το μέτρο αυτό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, τα άλλα κράτη-μέλη δεν αυξάνουν την παραγωγή όσο θα μπορούσαν, άρα διατηρείται μία ισορροπία όσον αφορά την παραγωγή της ζάχαρης. Δεν επηρεάζει η ισορροπία αυτή από το μέτρο αυτό της προαιρετικής δεδεμένη στήριξης. Και βέβαια υπήρξε μια μείωση της τιμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όντως δεν κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα ε, δημοφιλή για τις χώρες εκεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που εξηγούν αυτό. Το δεν υπάρχουν πλέον ε, οι ίσως όσον αφορά τη ζάχαρη και είχαμε και μια αύξηση στην παραγωγή τα τελευταία χρόνια η οποία παρατηρήθηκε κυρίως στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εφαρμόζουν την προαιρετική στεδεμένη στήριξη και στο 80% των χωρών που εφαρμόζουν την προαιρετική στεδεμένη στήριξη η παραγωγή της ζάχαρης μειώθηκε, δεν αυξήθηκε. Συνεπώς, δεν θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό της προαιρετικής στεδεμένης στήριξης έχει μια γενική αρνητική επίπτωση όπως υπόθηκε. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω, Λίπρο Πρόεδρος. Είπατε ότι υπάρχουν 11 χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν την προαιρετική στεδεμένη στήριξη. Πρέπει να πάρουν άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κάνουν αυτό ή προβλέπεται αυτόματα από την κοινή γεωργική πολιτική, έτσι δεν είναι. Ή πρέπει να απευθυνθούν σε εσά εκ των προτέρων και να πάρουν από εσά άδεια προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την προαιρετική στεδεμένη στήριξη. Πώ λειτουργεί το σύστημα. Δεν ξέρω ακριβώ πώ λειτουργεί για το σημείο αυτό η κοινή γεωργική πολιτική υπάρχει μια πρώτερη κοινοποίηση της απόφασης αυτής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας το ρωτώ αυτό ουσιαστικά γιατί θα ήθελα να ξέρω πώς έχει διαδικασία και πώς συνεργάζεται κυρίως με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, τη DG DEFCO δηλαδή, ή πώς συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Γιατί ξέρετε ότι στα πλαίσια της συνθήκης θα, θα πρέπει να μην εξετάζουμε μόνο την τεχνική πλευρά, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με το PCD, δηλαδή με τις πολιτικές όσον αφορά την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν μπορείτε σήμερα να μου δώσετε εσείς κάποια απάντηση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια με άλλους εργαζομένου με τους οποίους να μην έρχεστε αναγκαστικά σε επαφή. Θα ήταν πάντως ιδιαίτερα χρήσιμο για μας να γνωρίσουμε ακριβώς πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία και αν θέλετε και το όλο ιστορικό όσον αφορά τις επιδοτήσεις για την καλλιέργεια ζαχαρότευτων γιατί εδώ και 10 χρόνια μας απασχολεί η ιστορία αυτή και σίγουρα χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό και στα πλαίσια της προηγούμενης κοινή γεωρικής πολιτικής. Απάντηση. Δεν έχω κατά νου το σύνολο τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν ασχολούμαι ακριβώ με το ζήτημα αυτό. Προφανώ όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τι απαραίτητε πληροφορίε, άρα τα κράτη-μέλη κοινοποιούν σε κάποια φάση την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσουν την προαιρετική στεδεμένη στήριξη στον τομέα τη ζάχαρη. Επομένω, Έχουμε και μια ιδέα, μια εικόνα του αριθμού των κρατών μελών που θέλουν να εφαρμόσουν το μέτρο αυτό. Και επίση μας λένε σε ποιον τομέα θα το εφαρμόσουν και με τι προπολογισμό. Πάντως μπορούμε να σας δώσουμε και πιο συγκεκριμένε πληροφορίες. Ενδεχομένω ε, να έπρεπε να θέσουμε τουλάχιστον στην επόμενη συνεδρίασή μα το ερώτημα αυτό. πώ λειτουργεί στην πράξη το σύστημα πώς κοινοποιούν την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το μέτρο αυτό τα κράτη-μέλη, ποιες είναι οι εσωτερικές διεργασίε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς τελικά το μέτρο αυτό εφαρμόζεται. Κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ θα μπορούσε να μας απαντήσει. Μισελ Ντεκνούπ, λέγομαι κυρία Πρόεδρε, από πλευρά Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, τη μονάδα που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των τροφίμων, όπου ασχολούμεθα με προϊόντα όπω η ζάχαρη, ασχολούμεθα και με το ζήτημα αυτό. Είμαι δίπλα εδώ πέρα στο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη και αυτό αποτελεί και απόδειξη της στενής μας συνεργασίας. Θα θέλαμε να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό και χαιρόμαστε που διεξάγουμε τη συζήτηση αυτή γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε και την πλευρά των Ευρωβουλευτών Καθώ επίση και των χωρών ΑΚΕ, γιατί ακούσαμε εδώ πέρα δύο διαφορετικέ προσεγγίσεις τελικά. Όταν βρίσκεσαι λοιπόν στη μέση των δύο αυτών πλευρών και όταν πρέπει ουσιαστικά να εξασφαλίσει μια κάποια συνεκτικότητα και συνέπεια, τα πράγματα περιπλέκονται. Α μην τα περιπλέκουμε εμεί ακόμα περισσότερο, γιατί εν τέλει μην το ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο τη ανεπτυξιακής πολιτική ασχολούμεθα με όλου του εμπλεκόμενου πολιτισμού, πληθυσμού, με συγχωρείτε, που εμπλέκονται στου τομεί. Στου οποίου επικεντρωνόμαστε. Όταν ακούμε λοιπόν τα αριθμητικά αυτά δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, τασόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Βλέπουμε δηλαδή ότι όντω σε τελική ανάλυση είναι συνεκτική η πολιτική, αλλά από την άλλη βλέπουμε και την άποψη των χωρών ΑΚΕ, όπου εκεί συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να είμαστε και είμαστε σε συνεχή διάλογο με τις αρχές των χωρών αυτών. Έχετε τους αρμόδιους πρέσβεις και πρέπει να σας πω ότι όλοι οι συνάδελφοι από τις πρεσβείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλαμβάνονται του θέματος αυτού στις επαφές που έχουν με τις τοπικές αρχές και αν θεωρούμε ότι ε, στα πλαίσια της συμφωνίας περιλαμβάνεται και ο αγροτικός τομέας ή ο τομέας της ζάχαρης, τότε σίγουρα θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένε πολιτικές αλλά και συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να στηριχθούν οι χώρες αυτές που το έχουν ανάγκη. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι ε, αν η ζημία αυτή έχει αποτιμηθεί όπως ακούσαμε σε 20 εκατομμύρια ετησίως, πρέπει να σας πω ότι ε, το ποσό αυτό ουσιαστικά καλύπτεται από όλη τη χρηματοδοτική συνδρομή που πηγαίνει προς τις χώρες αυτές. Το θέμα λοιπόν είναι να καταφέρουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίξουμε τις χώρες αυτές που θέλουν να έχουν μια βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της ζάχαρης. Ελπίζω ότι κατάφερα τρόπον την να αποσαφηνίσω λίγο το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, λίγο λέει Πρόεδρος, αλλά όχι εντελώς. Είδα ότι ε, υπάρχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι που συναντιούνται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν απόψεις, αλλά αυτό δεν μας βοηθά απαραίτητα να έχουμε μια κοινή κατανόηση του ζητήματος. Δεν νομίζω ότι θέλουν άλλοι συναδελφοί το λόγο, άρα θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στον πρέσβη για να απαντήσει ενδεχομένως σε κάποιες ερωτήσεις ή για να αποσαφηνίσει κάποια σημεία. Και έπειτα ως Επιτροπή θα αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Ε, ε, Ευχαριστώ. Καταρχά, να ευχαριστώ τους δύο ευρωβουλευτέ που παρενέβησαν στο θέμα της Βραζιλίας και το θέμα της μεταρρύθμισης τη κοινής γεωργική πολιτική. Καλοδεχούμενα τα σχόλια. Γιατί συμπίπτουν ε, με κάποιες ανησυχίες που είχαμε από την πλευρά των χωρών και κυρία Πρόεδρε, οι εξολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την πλευρά τη της ομάδας ε, και έχουν διαφορές. Αναγνωρίζουμε ότι η στήριξη είναι από τα στοιχεία που επηρεάζουν τις αγορές. Και ότι υπάρχει μια αύξηση ευρωπαϊκής παραγωγής σε που δεν θα υπήρχε αυτό φυσικά επηρεάζει τις τιμές και γι' αυτό οι εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ζάχαρη από τις χώρες ε, ΑΚΕ επηρεάζεται. Ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα θέματα όταν υπάρχουν διαφορετικές ε, αξιολογήσεις είναι να συναντηθούμε, να βρεθούμε μαζί και να κάνουμε μια κοινή αξιολόγηση, να συζητήσουμε με μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουμε ε, είμαστε σε επικοινωνία και θεωρώ ότι μια καλή επικοινωνία με τους συναδέλφους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις ενδιαφέρομενες γενικές διευθύνσεις θα μας βοηθήσει να καταλήξουμε στο να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, με ανεξάρτητο τρόπο μια κοινή αξιολόγηση ώστε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο ίδιο έδαφος και από εκεί να προχωρήσουμε κυρία Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσα να ζητήσω να δω αν υπάρχει κάποιος από την πλευρά το χρονακέ που θα ήθελε να σχολιάσει. Παρακαλώ. Ε, σας παρακαλώ να είστε τον εαυτό σας. Πάτρικ Σαρντονέ εκπροσωπεί την βιομηχανία της ζάχαρης ε, της Δομινικανής Δημοκρατίας. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γρήγορος γίνεται. Είναι τιμή μου να μπορώ να μιλήσω εσά και στους συναδέλφου σα. Είμαι μπερδεμένο πάρα πολύ από την δήλωση τη Επιτροπή ότι είναι περιορισμένο το παιδί εφαρμογή των VCS των συμφωνιών στήριξη. αφορούν πάνω από 400.000 στρέμματα. 1,6 εκατομμύρια εκτάρια υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μου λέτε ότι 400.000 εκτάρια δεν είναι πολλά, τότε αυτό με εκπλήσει. Επίσης, 440 ευρώ ένα εκτάριο το εισόδημα είναι μεταξύ 2.000 ε, ε, και 2.200 ευρώ τα έστω από αυτά, από αυτά τα εκτάρια. Μιλάμε για 20% κέρδος. Είμαι πολλά χρόνια σε αυτό τον κλάδο, θεωρώ τον αυτό μου πυρογνώμονα. Είναι ένα ποσό το οποίο θα έχει ουσιαστική ε, επίδραση στον εφοδιασμό. Δεν μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν δύο με 3 εκατομμύρια τόνοι. Τώρα η ανάγκη της Ευρωπαϊκής είναι 18 εκατομμύρια τόνοι. Είναι μεγάλη διαφορά. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διπλασιάστηκαν σε 3 εκατομμύρια πέρσι. Καταστρέφουν την αγορά. Αυτές οι εξαγωγές καταστρέφουν ε, την περιοχή μας και την βιομηχανία μας. Το δεύτερο θέμα που με μπερδεύει και με Ευρωπαίος πολίτης είναι ότι ότι η δήλωση της Επιτροπής ότι τον Ιούνιο του 2018 η κατάργηση των ε, στηρίξεων θα έχει μικρή επίπτωση. 18.000 εκτάρια θα σταματήσουν να παράγουν ζαχαρότευτλα σε σχέση με τα 400.000 εκτάρια που λαμβάνουν ε, τις ε, επιδοτήσεις. Δεν ξέρουμε ποιος, ε, ποια νομοθεσία ισχύει εδώ τελικά. Η 1307 ή κάποια άλλη. Ε, ποιος είναι ο στόχος να υποστηρίξουμε την παραγωγή και να τη διατηρήσουμε. Αν κάνουμε λόγο για 400.000, αλλά τελικά μόνο 80.000 χρειάζονται ε, για να στηρίξουν την παραγωγή, τότε εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί ζητάτε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Μία με τρία εκατομμύρια τόνων που εξάγονται, μένουν επιδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τις εξαγωγικές επιδοτήσεις. Έχουμε όμως ε, πολιτική συνοχή για την ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και την Επιτροπή. Άρα θα προσπαθήσουμε από κοινού να βρούμε έναν τρόπο να το συντονίσουμε το θέμα αυτό και να το προχωρήσουμε. Ε, ίσως ζητήσουμε από την Επιτροπή να το διερευνήσει. Κάνουμε λόγο και για την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική. Παράλληλα, ίσω θα πρέπει επομένω να προτείνουμε τροπολογίε για την μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική πάνω στα θέματα αυτό. Κυρία Χόιμπουκ, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Θα προτείνει τροπολογίε. Θα το αφήσουμε εδώ για σήμερα. Θα ευχαριστήσω τον πρέσβη και την επιτροπή που ήταν παρούσα σήμερα το πρωί. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο το θέμα. Ε, το ξύσαμε επιφανειακά σήμερα, θα πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ καλύτερα όμω. Ευχαριστώ πολύ. And now, colleagues, moving to joint mode. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με την από κοινού συνεδρίαση με την Επιτροπή Ίντα